I αρχίσουμε γιατί περνάει η ώρα. Έχουμε ήδη χάσει ένα τέταρτο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σε ενημερώσω ότι υπάρχει ένα αίτημα από το Jens Kair να αλλάξουμε το σημείο 10 τη σειρά του το σημείο 10 που αφορά τις περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές. Έχουμε μια πρόταση από το συνάδελφό μας να το συζητήσουμε μετά τις 5 γιατί δεν μπορεί να έρθει νωρίτερα. Αν συμφωνείτε λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για τα σημεία 12 και έως 16 θα περάσουν μία ώρα νωρίτερα και θα ξεκινήσουμε γύρω στις 3.30. Αν συμφωνείτε, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σας θυμίζω επίσης ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανή στο ίντερνετ. και ο χρόνος που προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη είναι βεβαίω πάντα ενδεικτικό γιατί ε, για απρόβλεπτους λόγους ορισμένε φορές χρειάζεται να μεταβληθούν ε, οι χρόνοι συζήτηση. Περνάμε στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 17 η 18 δεκεμβριου Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα, έχουν διανεμηθεί, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί στο τέλος της ε, συνεδρίασής μας, εάν δεν εγερθούν αντιρρήσεις. Τρία, ανακοινώσει της Προέδρου. Δεν έχω. Οπότε περνάμε στο σημείο 4, που είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης καλέσαμε και τον εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειών για να κάνουμε μία λοιπόν ανταλλαγή απόψεων για τις νέες περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, τις κατευθυντήρες γραμμές για το θέμα αυτό. Καλώ λοιπόν τον πρώτο μας ομιλητή, Χέρτ Γιάν Κόπμαν, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για τις κρατικές ενισχύσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ακούσουμε τον Νίκολας Μάρτσιν της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειών. Παρακαλώ, Χερδιάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Χιούμπνερ για την εισαγωγή σας και καλημέρα. Ξεκινώντας ε, να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ στην Επιτροπή σας για να σας παρουσιάσω σύντομα τον τρόπο σκέψης μας για τις ε, κατευθυντήρες γραμμές, για τις ε, περιφερειακές ενισχύσεις και να έχουμε ένα διάλογο με το Κοινοβούλιο. Ο επίτροπο μου, αντιπρόεδρο Αλμούνια, θα ήθελε να παρευρίσκεται, αλλά δυστυχώς δεν είχε δυνατότητα σήμερα. Υπογραμμίζω ωστόσο ότι είναι πάντα διθέσιμο για να συζητήσει μαζί σα για το θέμα αυτό, γιατί η σημαντική του, συμβολή του Κοινοβουλίου είναι εξόχως ενδιαφέρουσα για μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις είναι ένα στοιχείο μιας πολύ ευρύτερης μεταρρύθμισης των κρατικών ενισχύσεων που καλύπτει όλους τους κανόνες και τους διαδικαστικούς για τον έλεγχο αυτών των επιδοτήσεων στην Ένωση. Το πακέτο αυτό που το αποκαλούμε εξυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων, ΣΑΜ, έχει τρεις στόχους. Ο πιο σημαντικός είναι να ενθαρρύνουμε την οικονομική ανάπτυξη και να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, στοχεύουμε στη διασφάλιση της μείωσης της γραφειοκρατίας και επίσης η Επιτροπή έχει στόχο να επικεντρώσει, να εστιάσει την προσοχή της στις κυριότερες ενέργειες που αφορούν την εσωτερική αγορά. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Τα αναφέρω γιατί οι περισσότερες επιπτώσεις ε, των αλλαγών στις κρατικές ενισχύσεις, επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής, θα προκληθούν από πολλές μεταρρυθμίσεις του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων που θα εισαγάγουμε. Οι περιφερειακές κατευθυντήρες γραμμές είναι μόνο ένα τμήμα αυτών των αλλαγών. Σημαντικό αυτό. Γιατί έχω ακούσει ανησυχίες που όμως πιστεύω ότι αντιμετωπίζονται αν εξετάσουμε και κάποιες άλλες πλευρές αυτού του πακέτου αλλαγών. Βλέπετε εδώ ένα πίνακα που ίσως να είναι λίγο δυσνόητος, αλλά να σας τον παρουσιάσω. Τι βλέπετε σε αυτό τον πίνακα? Βλέπετε ότι κατά την περίοδο την τρέχουσα προγραμματισμού η πολιτική συνοχής ήταν ύψους 375 εκατομμυρίων. Είναι λοιπόν τμήμα των ευρύτερων δαπανών για την περιφερειακή πολιτική συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών πόρων που είναι περίπου 5 δις. Από αυτά τα ποσά μόνο περίπου 20%, 70 με 80 δις ε, εκατομμύρια είναι κρατικές ενισχύσεις. Ο μεγαλύτερος λοιπόν το μεγαλύτερο τμήμα λοιπόν ε, της ε, πολιτικής συνοχής δεν είναι χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή. Τι ε, όργανα χρησιμοποιούμε τώρα για να ελέγξουμε την, τις κρατικές ενισχύσεις, τις περιφερειακές ενισχύσεις. Θα δείτε ότι η πρώτη κάθετη στήλη καλύπτει μόνο ένα μικρό ποσοστό των δαπανών για την πολιτική συνοχή που θεωρούμε ότι είναι ενισχύσει. Θεωρούμε ότι είναι λιγότερο από, το, από τα 70-80 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τα δύο τρίτα είναι υπό άλλε κατευθυντήρε γραμμέ που θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικές για τον έλεγχο των ενισχύσεων. Αφορούν λοιπόν την ε, πολιτική συνοχή ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν οι κατευθύνσεις για την έρευνα και την καινοτομία και την περιβαλλοντική ενίσχυση. Και έχουμε και άλλες ενισχύσεις που όμως αφορούν ένα μικρότερο ποσοστό του ποσού. Ναι μεν λοιπόν είναι σημαντική αυτή η συζήτηση για τις περιφερειακές ενισχύσεις αλλά αφορά ένα μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης και τώρα αλλά και στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εξίσου σημαντικό, πιστεύω, είναι αυτό που αφορά τον ορισμό της περιφερειακής ενίσχυσης, που είπα πως είναι περίπου το 1 τρίτο των ενισχύσεων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Από αυτό το 1 τρίτο, περίπου το 60% το διαχειρίζεται ενεργά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις λεγόμενες ενημερώσεις όπου η Κομισιόν εξετάζει την συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων μέτρων αλλά περίπου 40% εξαιρείται. Δεν χρειάζεται να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον κάποιες βασικές προϋποθέσεις στηρούνται. Βασικό μου λοιπόν ε, σημείο είναι η έκκληση που κάνω προς την Επιτροπή σας να δει ευρύτερα τις ε, κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και να μην θεωρήσει ότι οι περιφερειακές κατευθύντηρες γραμμές ε, για τις κρατικές ενισχύσεις είναι το βασικό στοιχείο και το μόνο. Ένα στόχος αυτής της προσπάθειας εξχρονισμού που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Αυτό αντανακλάται σε όλες τις κατευθύντηρες γραμμές που τροποποιούμε προσπαθώντας ε, να έχουν πιο ουσιαστικές επιπτώσεις οι ενισχύσεις μας. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι ποσοστό, τι αποτέλεσμα μάλλον ε, κινητοποίησης και άλλων πόρων έχουν οι ενισχύσεις μας. Δηλαδή να αποδίδουμε την ενίσχυση εκεί που θα έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Βεβαίως έχουμε ήδη μεγάλη πείρα από τη χρήση των πόρων μας στο παρελθόν και σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι κάποιες χρηματοδοτήσεις δεν δαπανώνται όσο σωστά και αποτελεσματικά και σοφρόνος θα έπρεπε. Αυτό μας ανησυχεί βεβαίως, γιατί δεν είναι σκόπιμο να δώσουμε για παράδειγμα υψηλέ ενισχύσει επιχειρήσει που διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό τη στην εσωτερική αγορά. Αλλά βεβαίω πρέπει και εσά να σε ενδιαφέρει, διότι οι περιορισμένοι πόροι για τη συνοχή πρέπει να δαπανώνται αποτελεσματικά. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη χρήση των πόρων για τη συνοχή. Είναι κοινό λοιπόν ο στόχο μα. Θα πρέπει οι ενισχύσει αυτέ να είναι αποτελεσματικέ. Και τι προτείνουμε σε αυτέ τι νέε καθευθύντηρε γραμμέ είναι να τονίσουμε πολύ περισσότερο την αποτελεσματικότητα λοιπόν των ε, ενισχύσεών μα. Βεβαίω έχουν υπάρξει κάποιε διαφωνίε για κάποιο σημείο. Και συγκεκριμένα για τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαγορεύουν τις ενισχύσεις σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στις ε, περιοχές της λεγόμενες τύπου C. Είναι πιο αναπτυγμένες όπου 75-90% του κατακεφαλήν σε σχέση με το μέσον όρο της Ένωσης. Αυτές οι περιοχές είναι περιοχές στις οποίες, για τις οποίες τα κράτη-μέλη έχουν ε, ευρεία δυνατότητα καθορισμού. Και η έρευνα που έχουμε κάνει και από τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής καταδεικνύουν ότι οι επιδοτήσεις που δίνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές δεν αλλάζει στην ουσία τη συμπεριφορά αυτών των μεγάλων εταιριών. Δηλαδή συνεχίζουν να έχουν τις ίδιες δραστηριότητε δαπανούν περίπου το ίδιο ποσοστό πόρων που θα δαπανούσαν και χωρίς τις ενισχύσεις. Και αυτό μας ανησυχεί, διότι αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν διαμεθοριακή δραστηριότητα και άρα είναι πιθανόν να λαμβάνουν ε, αδικαιολόγητα υψηλά ποσά επιδοτήσεων. Έχουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό, αναλυτικά και ε, διαχειριζόμενοι διάφορες ε, επιδοτήσεις. Βλέπουμε διάφορες επιχειρήσεις που ε, κοιτάνε σε πολλές χώρες της Ευρώπης να δούνε πού μπορούν να πάρουν επιδοτήσεις. Θα δημοσιεύσουμε σύντομα τις δέκα πρώτες μεγάλες επιχειρήσεις από πλευράς λήψης κρατικών περιφερειακών ενισχύσεων και θα εκπλαγείτε όταν θα διαπιστώσετε ότι είναι οι ίδιες επιχειρήσεις, πολύ συχνά αυτοκινητοβιομηχανίες που λαμβάνουν από διάφορες κυβερνήσεις ενισχύσεις, συνήθως για τα ίδια προγράμματα, τις ίδιες δραστηριότητες. Στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι να αντισταθμίσουμε την, να αντισταθμίσουμε την ε, πολιτική μας ούτως ώστε να μην προκαλεί ε, στρεβλώσει ανταγωνισμό. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει οι είναι πολύ πιο χρήσιμες, ε, είναι πολύ πιο χρήσιμο να λαμβάνουν επιδοτήσει από τι μεγάλε. Βεβαίω και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα. Αλλά είπα ότι η ενισχύση προ αυτέ τι μεγάλε επιχειρήσει δεν ενισχύει περαιτέρω δραστηριότητε του. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο αλλά δύο σημαντικές επιφυλάξεις σχέση με αυτό. Όπως βλέπετε και εδώ στη διαφάνεια, υπάρχουν και άλλες κατευθύντηρες γραμμές που επιτρέπουν να χορηγούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις ε, επιδοτήσεις για έρευνα, καινοτομία και περιβαλλοντική επίσης βοήθεια για θέματα όπως ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Φυσικά αυτό θα συνεχίσει να είναι επιτρεπτό σε όλες τις χώρες και όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. Δεν πρόκειται λοιπόν να απαγορεύσουμε τις ενισχύσεις της μεγάλης επιχειρήσης. Θα περιορίσουμε όμως το εύρος αυτών των ενισχύσεων. Και αυτό συμφωνεί και με τις ευρύτερες προτάσεις κανονισμών για την περιφερειακή πολιτική. Το δεύτερο. Μετά από συζητήσεις για το θέμα αυτό, ο Αντιπρόεδρος Αλμούνια είπε ότι θα ήταν ανοιχτή η Επιτροπή να διερευνήσει μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς τις συνθήκες υπό τις, επίες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να υπάρξουν στοχευμένες εξαιρέσεις προς τον κανόνα αυτό για να γίνουν επενδύσεις όπου η προστιθέμενη αξία ή η προσθετικότητα μπορεί να αποδειχθούν. Δεν ε, κλείνουμε λοιπόν εντελώς την πόρτα σε σχέση με αυτό, αλλά θεωρούμε ότι επί της αρχής έχει σημασία να εφαρμοστεί αυτή η νέα πολιτική. Και όπως είπα εμένουμε να υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ένα τελικό σημείο είναι ακόμη περισσότερη προσοχή στις αρχές της διαφάνειας και μελέτης επιπτώσεων και αποτελεσματικότητας. Είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή εφαρμογή αυτής της πολιτικής να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση για το ποιοι λαμβάνουν ενισχύσει, ποιοι είναι οι στόχοι, όλα αυτά να είναι δημοσίως γνωστά, να μπορεί να τα διερευνά η κοινωνία των πολιτών και οι εκλεγμένοι φυσικά εκπρόσωποι όπως εσείς είναι οι κανόνες λοιπόν, θα απαιτούν τα στοιχεία αυτά να δημοσιεύονται με τρόπο που να είναι προσβάσιμο σε όλους. Δεύτερον, για σημαντικές δαπάνες όπου έχουμε τα λιγότερα γενικά προγράμματα, schemes, μας ενδιαφέρει αυτά τα γενικά προγράμματα να αποτιμώνται τακτικά για να διαπιστώνεται η σωστή χρήση των χρηματοδοτήσεων. Και αυτή η πρόταση λοιπόν θα υποβληθεί ούτω ώστε όταν είναι πολύ μεγάλα τα προγράμματα να αποτιμώνται ούτω ώστε όλοι να εξάγουμε διδάγματα από την πείρα χρήσης αυτών των μεγάλων διαστάσεων προγραμμάτων. Αυτά είναι οι κυριότεροι στόχοι, οι κυριότερες αλλαγές. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά ίσως να επανέλθουμε στις ερωτήσεις. Πρόεδρος, ναι, εντάξει. Να ζητήσω τώρα τον Νίκολας Μάρτιν ε, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας δώσω τις ε, προοπτικές που εξετάσαμε σε σχέση με την ε, έρευνα που κάναμε για τον εξεχρονισμό των κρατικών ε, ενισχύσεων και την, την εκπόνηση των κατευθυντήριων γραμμών της περιφερειακής πολιτικής. υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα σε ένα τομέα όπου υπάρχουν μεγάλες αλληλοεπιδράσεις γιατί η πολιτική συνοχής ε, υπάγεται στους κανόνες ε, της ε, κρατικής ενίσχυσης. Εμείς είδαμε με τη δική μας προοπτική τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η απλούστευση γιατί μία από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να απλουστεύσει την παροχή των ε, ποσών των ταμείων και να υπάρχει μία ε, ε, συνεκτικότητα σε αυτά τα σχέδια και λαμβάνουμε υπόψη μας διάφορα στοιχεία γι' αυτό. Είναι λοιπόν η διαπίστευση ένα πολύ σημαντικό σημείο για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν είναι φορτίο γραφειοκρατικό επιπρόσθετο απαραίτητα ε, ούτε υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιάμεσοι που δυσχεραίνουν τη διαδικασία. Ε, γίνεται εδώ λόγος για μια πολιτική η οποία να είναι συνεπής προς τον εαυτό της δηλαδή προς τους στόχους που έχει θεσπίσει ε, ανάλογα με τα διάφορα μέρη που ασχολούνται με αυτή την πολιτική. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καθοριστεί αυτή η πολιτική, θα επανέλθω από αυτού. Και επίσης είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας και των στόχων που έχουμε για το πακέτο της πολιτικής συνοχής που έχει μια συνολική αποτελεσματικότητα για τη χρήση των διατεθειμένων ποσών ε, Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεκτικότητα σε πιο λεπτομεριακό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές των κατευθυντηρίων γραμμών της περιφερειακής πολιτικής για τους οποίες έχουμε και τους ανάλογους χάρτες. Έχουμε εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ ε, των περιφερειών δηλαδή μια απόδειξη της ε, ε, συνοχής της περιφερειακής πολιτικής που είναι και διασυνοριακή. Έτσι η απλούστευση έχει σαν στόχο τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν αφορά μόνο τις κατευθυντήριες γραμμές αλλά όπως είπε και ο Γκέρτ Γιάν Κούπμαν ε, είναι ένα θέμα αλληλοεπίδρασης μεταξύ της κρατικής πολιτικής ενισχύσεων και της περιφερειακής πολιτικής. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις κατευθυντήριες γραμμές γιατί εδώ φαίνεται η βλάβη που υπάρχει σε σχέση με την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχουν οι χάρτες οι οποίοι μας δείχνουν ότι τίθεται ένα θέμα συνοχής συγκεκριμένης για την εφαρμογή της ε, περιφερειακής πολιτικής πώς γίνεται η διανομή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί. Τώρα για την ίδια τη διαδικασία έχουμε μία φάση καταρχήν ε, ε, διαβουλεύσεων και οι γενικές διευθύνσεις οι αντίστοιχες ήταν πολύ δραστήριες εξετάζουν τη διαδικασία το πώς έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα προαναφερθέντα θέματα ε, και έχουμε μια διαδικασία την οποία ακολουθούμε και υπάρχει ένα κείμενο που έχει αποσταλεί σε όλους για τη διαβούλευση όπου εκφράζει διάφορες ανησυχίες παραδείγματος χάρη για το θέμα της ε, υποστήριξης αν είναι ε, κατάλληλη και επαρκής η υποστήριξη ε, κατά κατηγορία και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην προσέγγιση της κρατικής ενίσχυσης. Όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν τα προβλήματα γιατί έχει ληφθεί η απόφαση να υποστηριχθούν ορισμένα προγράμματα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι υπάρχει ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα της απλούστευσης ε, και υπάρχει και η, η, ειδική μεταχείριση της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τις περιφέρειες. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να ε, έχουμε αποφύγει τις διάφορες ανομαλίες και τις διάφορες ασυνέπειες στην εφαρμογή των κατευθυντηριών γραμμών. Αλλά η πολύ καλή ενίσχυση της ε, συνέργειας με τις ε, κρατικές πολιτικές είναι κάτι που θα μας βοηθήσει περαιτέρω. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι χάρτες που εκπονήσαμε για να καθορίσουμε τις κατηγορίες των περιφερειών για την πολιτική συνοχή, η οποία θα χρησιμοποιήσει σαν σημεία αναφορά στα δεδομένα από το 2007 στο 2009 και ε, την αναφορά ε, σε μία περίοδο που θα είναι περίοδος αναφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή 2009 με 2010 ε, και θα δούμε τα διαθέσιμα στοιχεία όταν θα προκύπτει κάποιο σημείο που θα χρειάζεται ενδελεχή συζήτηση και πρέπει να δούμε ότι έχουμε ε, κάνει ορισμένες προσωμιώσεις και μπορούμε να ε, έχουμε στη συνέχεια συγκρίσεις όταν πρόκειται να αναλάβουμε συγκεκριμένη ε, δράση για να αποφύγουμε τις οποιασδήποτε ανομαλίες. Για το θέμα τώρα των μεγάλων επιχειρήσεων υπάρχει εδώ ένα τεράστιο ένα πεδίο όπου υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες με τα προβλήματα τα οποία είχαμε συζητήσει για τις κρατικές ενισχύσεις πολλές φορές εδώ είχαμε συζητήσει με προτάσεις της Επιτροπής ε, και υπάρχει μια ομοιότητα με τα στοιχεία που μας έφεραν οι συνάδελφοί μας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, τις αξιολογήσεις που γίνονται και φαίνεται ότι πολλές φορές δίνεται μια υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλη στις μεγάλες επιχειρήσεις και πάντα είναι πιο αποτελεσματική, έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η ενίσχυση που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι αυτή που δίδεται στις πιο μεγάλες. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο για την ώρα βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στον τρίλογο που γίνεται μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου και γι' αυτό για την ώρα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε εκπονήσει μια τελική θέση ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια προσέγγιση η οποία χαρακτηρίζεται καταρχήν από ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να διατηρηθούν. Βεβαίως να περιορίσουμε ε, την ατζέντα που έχουμε για τον καθορισμό των ε, κατηγοριών και των τιμών. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές που έχουν ε, θέματα με την ανανέωση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της ενέργειας και μια πιο ειδική στάση ως προς την ανάπτυξη η οποία είναι αναγκαία και απαραίτητη. Αυτά τα θέματα τα οποία ανάφερα στην αρχή λοιπόν φαίνεται να μην έχουν αλλάξει πάρα πολύ γιατί δεν προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος ε, προβληματισμός για αυτά. Ε, θα δούμε τώρα τις εσωτερικές διαδικασίες καλύτερα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το ότι θα διατηρήσουμε ε, όλη αυτή τη συνεκτικότητα που είναι αναγκαία για την τελική ε, μορφή που θα λάβουν οι κατευθυντήριες γραμμές όταν εγκριθούν από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Ζαμπόλ Ντερανό που είναι από την Επιτροπή Περιφερειών να είναι εισηγητής να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση είμαι εδώ ανάμεσά σας. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκλησή σας για να σας πω ποια είναι η άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών για τις κατευθύνες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 2014-2020. Εξ ονόματο της Επιτροπής Περιφών θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας αυτή. Αυτές οι ενισχύσεις επειδή ακριβώς παίζουν ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη είναι μέρος των εξαιρέσεων των απαγορεύσεων που υπάρχουν που είναι γεγραμμένες στην ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και για τη δημιουργία επιχειρήσεων και για τα έξοδα λειτουργίας για τη σύσταση επιχειρήσεων κλπ. Και εκεί που η ιδιωτική επιχειρηματικότητα αποκλείει την ε, ενεργοποίησή της, η και γι' αυτό ακριβώς ε, τώρα τελευταία ομόφωνα εγκρίθηκε μια κοινή γνώμη για το μέλλον αυτών των ενισχύσεων. Ε, και ο στόχος ποιος ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνουμε ώστε να μην περιοριστούν αυτές οι δυνατότητες δημόσιας παρέμβασης υπέρ των επιχειρήσεων και αντίθετα να συνεχιστούν και αποτεσματικό να υποστηρίζουν τις διάφορες περιφέρειες για να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει από την οικονομική ανάπτυξη και στο κοινωνικό πλαίσιο, το κοινωνικό, οικονομικό, Αυτές ε, οι υπηρεσίες κατά την άποψή μας όλο και περισσότερο είναι απαραίτητες. Σαν μέλος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη ακριβώς βέβαια ε, δείχνεται ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτό το θέμα και αυτές οι κρατικές ενισχύσεις είναι αρμοδιότητες αποκλειστικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αλλά τουλάχιστον και επειδή έχουν στόχο τις περιφέρειες, απαραίτητο κατά την απόψή μου είναι ε, εμείς ε, οι εκλεγμένοι εκεί και εσείς να μπορέσετε να εκφραστείτε και να μπορέσουμε να εκφραστούμε για να παίξουμε τον ρόλο που πρέπει στις όλες διαπραγματεύσεις. 14 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε, δημοσίευσε τις νέες κατευθυντικές γραμμές με μια δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή Περιφερειών είναι η πρώτη που εξέφρασε την απόψή της και Αποφελούμε σήμερα από την πρόσκλησή σα για να σε ενθαρρύνω και εσεί να εκφράσετε την απόψή σα πάνω στο θέμα αυτό. Και η Επιτροπή Περιφερειών είχε γνωμοδοτήσει με πρωτοβουλία τη ε, και να δείξει ακριβώ και στην Επιτροπή το ενδιαφέρον που είχε ο χώρο αυτό με το θέμα αυτό και από το ξεκίνημα των συζητήσεων στην Επιτροπή Περιφερειών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι προχωρήσαμε κάπως σχετικά με το κείμενο και στην τελευταία συνάντησή μας στην Ολομέλεια ο Ιωκή Μαλμούνια ο Επίτροπος ακριβώς άλλαξε την αποφασή του για τη μείωση του σνού του πληθυσμού καλύπτεται από τις ενισχύσεις αυτές ήταν ένα σχέδιο ακριβώς αρχικό το οποίο εγκαταλείφθηκε και αυτό μας ικανοποιεί. Πρόκειται για ένα πρώτο νέο για τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Αλλασμένα από αυτά που έχουμε ζητήσει προς στιγμή να αποτελούν πάντα νεκρό γράμμα και θα πρέπει να επιμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Και υπάρχει ο περιορισμό για την χωρίς αυτής της βοήθειας. Αλλά αυτός ο περιορισμό θα ήταν λάθος και στα πλαίσια αυτά μιας κρίσης στην οποία ζούμε θα είχε ιδιαίτερη αρνητικές επιπτώσεις ε, πάνω σε πληθυσμό που ήδη υποφέρει και με τη βοήθεια αυτή θα μπορέσουμε να πετύχουμε ε, κοινωνική, οικονομική σύγκληση, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε μια νομισμένη ανάπτυξη των διαφορών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να δούμε τις απαιτήσει τώρα της Επιτροπής μας Περιφερειών στα πλαίσια αυτά τα οποία μόλις σας εξέθεσα. Η πρώτη απέτηση είναι αυτή η βοήθεια και με μια συνοχή όλα αυτά συνδυαστούν με την, με την ε, πολιτική συνοχή. Μιλάμε για συνοχή ακριβώς έχει σημασία και γι' αυτό θα πρέπει να αναγνωστεί το καθεστώς ε, με το βεταβατικό αυτό των περιφερειών και στο σχεδιασμό των περιφερειών που θα αφορά αυτή η σύγκληση. Και είναι μια μετάβαση ιστορική μπορούμε να πούμε, αλλά και το αντίθετο και ε, υπάρχει μια διάκριση που δεν δικαιολογείται για περιφέρειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες. Είναι εκείνε που έχουν φύγει από τη σύγκληση και από την ανταγωνιστικότητα και που πραγματικά είναι κάτω από το 80% του ΕΠ, άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζονται εξίσου αυτές οι δύο κατηγορίες περιφερειών και θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Και οι περιφέρειες που είναι στα πλαίσια της, του ανταγωνισμού δεν μπορούν εύκολα να καλύψουν την το έδαφος. Και αυτό που θα θέλαμε είναι να αποφύγουμε την ε, Αυτέ τι κριτικέ κριτικές βέβαια, αλλά θέλουμε από την Επιτροπή με συνοχή πάντα με τον κανονισμό για τα ορτικά ταμείο να έχουμε μια αντίθετη με την, με την κατάσταση πολιτική και με ορισμένε συνθήκε dumping που επικρατούν σε διάφορε επιχειρήσει. Δεν καταλαβαίνουμε την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει τι ενισχύσει εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 250 εργαζόμενοι και που ακριβώς θεωρούνται σαν μεγάλες επιχειρήσεις, άδικα όμως, σαν να είναι πολυεθνικές. Αυτό το αναφέρατε προηγουμένως και νομίζουμε ότι είναι σημαντικό. Αυτές οι επιχειρήσεις κυρίε και κύριοι είναι τοπικές επιχειρήσεις και οικογενειακού τύπου πολλές φορές και ουσιαστικά είναι κυτρία δύναμη στον χώρο αυτό και ε, αφορούν πολλές θέσεις εργασίας. Ζητάμε από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την απόψή της ε, γι' αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι 250 εργαζόμενοι ενώ άλλες ανταγωνιστικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ορισμός τους είναι πολύ πιο ευέλικτος ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Μηχανίας εδώ διακυβεύεται πάνω σε αυτό το θέμα η Επιτροπή Περιφέρειων σήμερα κάτι άλλο. Να σας πω ότι προσέχει ιδιαίτερα για αυτή τη χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού χαρακτήρα ενδιαφέροντος και ζητάμε από την Επιτροπή να εξαιρέσει αυτή τη βοήθεια και που έχουν σχέση με την άμεση ενίσχυση του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευαίσθητο θέμα για το μέλλον αυτών των υπηρεσιών. Κάτι ακόμα. Παρακαλώ Προσέξτε, το ελάχιστο κατόφλι 200.000 ευρώ σήμερα, το γνωρίζετε, θα θέλαμε να έρθει στις 500.000 ευρώ για μια αποτελεσματικότερη παρέμβαση. Κάτι ακόμα. Θα πρέπει να συλλογιστούμε κατάλληλα για το πόσο πληθυσμό θα πρέπει να αφορά αυτή η περιοχή και ξεχνάμε πολλές φορές ότι υπάρχουν δεσμενείς συνθήκες και χρειάζονται ειδική κρατική ενίσχυση σε αυτές τις περιοχές. Τελευταίες διεκδικήσεις μας, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικές. Ε, Ακριβώ επειδή αυτέ οι κρατικέ ενισχύσει πάνε σε περιφέρειε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ειδικό χαρακτήρα διαφόρων περιφερειών και θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το ειδικό καθεστώς στις ε, υπερπεριφερειακές περιοχές ε, αλλά και να διαφέρουμε ιδιαίτερα εκείνες που έχουν ε, γεωγραφικά και αγροτικές περιοχές ή να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες είτε είναι επειδή είναι και νησιωτικές και θα πρέπει να ανησυχούμε γιατί από τη στιγμή που θα ε, επιληφθεί της καταστάσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουν να βοηθούν σε τοπικό επίπεδο. Είναι τεχνικό με το θέμα και επηρεάζει για την κατάσταση ανάλογα βέβαια με τον ειδικό χαρακτήρα κάθε περιφέρειας, κάθε περιοχής. Ε, μας αφορά όλους όμως αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τις προσπαθήσει, να συμμαχίσουμε και ε, χαίρομαι που θα ασχοληθείτε με το θέμα αυτό και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω στα ενδεχόμενα ερωτήματά σας και σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή που μου αφιερώσατε. Ε, Κρέλ, η κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπήρξε κάποια ανησυχία όταν δημοσιεύθηκε το έγγραφο της Επιτροπής, έντονη μάλιστα θα έλεγα, διότι θεωρήθηκε ότι δύο τομείς πολιτικής που σχετίζονται δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Κατά τη συνεργασία μας ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να διαπιστώνουμε εάν αυτά τα οποία εγκρίνουμε για την πολιτική συνοχή δεν θίγουν την πολιτική ανταγωνισμού. Είχα πολλές ανησυχίες, αλλά από τις ε, εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις που έγιναν κάπως έχω καθησυχάσει. Διότι η κατηγοριοποίηση των περιοχών ε, μου είχε δοθεί η εντύπωση ότι δεν ε, συμβιβάζεται με αυτά που αποφασίζει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, όλο το θέμα της απλοποίηση θα μπορούσαμε να το αφήσουμε κατά μέρο. Δεν θα είχε καμία επίπτωση οποιαδήποτε προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιες αντιφάσεις. Παρ' όλα αυτά, η συνεργασία για τον ανταγωνισμό είναι σημαντική μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Βεβαίως η συνοχή είναι θέμα συναπόφασης. Βεβαίως για τις ε, ε, μεγάλες επιχειρήσεις πολλές φορές η Κομισιόν έχει άλλη θέση από τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν ακόμη και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν τα 60 έως 80 δις ευρώ που αναφέρατε κύριε Κόμμαν ίσως να φαίνονται λίγα Μπορεί να μην είναι πρόβλημα για τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά είναι πρόβλημα για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές που είναι στην ενδιάμεση κατηγορία. Γιατί εδώ το τμήμα των ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγάλες είναι μεγαλύτερο. Γιατί έχουμε μόνο τρεις ή τέσσερις προτεραιότητες τις οποίες όλες πρέπει να εξυπηρετήσουμε με τις ε, επιδοτήσεις της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια συγκέντρωσης των πόρων μας. Και στο παρελθόν είχαμε πάντα και το εξής πρόβλημα. Συχνά. Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, πολύ συχνά οι επιχειρήσεις μετα... μεταφέρονται από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Μετεγκαθίστανται. Και βεβαίως εάν μία επιχείρηση θέλει να μετακινηθεί έχει μεγάλη σημασία να μην δυσχεραίνεται με αυτόν τον τρόπο η ε, κατάσταση της αρχικής της ε, περιοχής εγκατάστασης. Αυτές οι διαφορές λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού Δηλαδή να μην μετακινούνται οι επιχειρήσεις μόνο και μόνο για να πάνε να πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις σε κάποια άλλη περιφέρεια. Πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή τι κανόνες πρέπει να εκπονήσουμε για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ Κωνσταντς. Παρακαλώ όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις να το δηλώσουν γιατί ήδη έχουν ζητήσει το λόγο 11 και θα ήθελα να κλείσω τον κατάλογο. Οπότε παρακαλώ να είμαστε και πολύ σύντομοι όταν θα υποβάλουμε ερωτήσεις. Ο κύριος Φανίστελ Ευχαριστώ. το πιο σημαντικό. Είμαστε σε φάση ε, κοινή ε, νομοθετικής ε, αρμοδιότητας. Η πολιτική συνοχής θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και τώρα που διαπιστώνουμε ότι η Κομισιόν έχει κάνει προτάσεις που διαφέρουν από την παρούσα περίοδο χρηματοδότησης αυτά προκαλούν μια συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα ανταλλάσσουμε πληροφόρηση αλλά δεν επαρκεί θα πρέπει να είναι όμως πιο ε, δομημένη αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε και μια έκθεση σας παρακαλώ λοιπόν να μας διευκρινίσετε τι βήματα θα αναλάβετε και ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει πολύ σωστά διατυπωμένες ερωτήσεις για την Ολομέλεια. Πρέπει να δούμε τι περιοχές, πώς ορίζονται οι περιοχές. Ε, λαμβάνουμε υπόψη την πυκνότητα του πληθυσμού. Και αυτό που είπε και η Κωνσταντς για τα θέματα μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων. Ξέρουμε πόσο μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος μας. Πρέπει να θέσουμε πολιτικά στο κατάλληλο επίπεδο το θέμα αυτό. Ξέρω ότι η Κομισιόν παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά ίσως πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να πάμε λίγο παραπέρα. Ο Βίκτορ Μποστινάρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σκόπιμη γιατί πρώτη φορά συζητάμε τις κρατικές ενισχύσεις και την συνοχή ενώ συζητάμε για το μέλλον της Ευρώπης. Τι ρόλο θέλουμε να έχει στην ανάπτυξη της οικονομίας η Ευρώπη στο μέλλον, πώς θα επηρεάσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Διότι κάποια δόγματα που υιοθετούσαμε μέχρι πρόσφατα τυφλά έχουν κρίση. Ένα από τα βασικότερα ε, δόγματα ήταν ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι βλακώδεις και κακές ενώ οι ιδιωτικές είναι υπανάκια και εξορισμού σωστές. Τώρα βλέπουμε ότι πολλές μελέτες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ, στο Καναδά, την Ευρώπη αποδεικνύουν ότι εάν οι κρατικές ενισχύσεις ε, τύχουν σωστής διαχείρισης μπορούν να βοηθήσουν όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Δεύτερον, κατασκευαστικός τομέας κατά του τριτογενούς Πρόσφατα μας είπαν ορισμένα πράγματα, αλλά τώρα λόγω της κρίσης δεν βλέπουμε να ισχύουν. Οι χώρες λοιπόν που είχαν, που έχουν ε, ευρύ κατασκευαστικό τομέα, τα πήγαν καλύτερα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης από όσε ε, βασίζονταν κυρίως στις υπηρεσίες. Γερμανία σε σχέση με Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Ουγγαρία ή άλλοι όπου υπήρξε τεράστια από αποβιομηχάνηση, ενώ άλλες χώρες, όπως η Κίνα, τα πάνε καλύτερα. Τρίτο δόγμα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μετεγκαθίσταντο στο όνομα του κέρδους. Αλλά τι κάνουμε, εξάγουμε την τεχνογνωσία μας και εισάγουμε τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα και αλλού. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πολιτική αντιμετώπιση των μετεκαταστάσεων. Διότι ξέρετε ότι αν δεν το κάνουμε θα υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις Μιτάλ, Φλωράνζ, ε, Χαλιβουργία στην ε, Ρουμανία και το Λουξεμβούργο που κλείσανε. Θα πρέπει λοιπόν και βεβαίως ε, και στην Ιταλία υπήρξε πρόβλημα με τη Χαλιβουργία. Άλλο δόγμα. Το μικρό είναι ναι, μπορεί το μικρό να είναι γλυκό, αλλά κατά τη διάρκεια της κρίσης καταρρίφθηκε και αυτό το δόγμα. Δεν ισχύει τουλάχιστον όπως θεωρούσαμε ότι ίσχυε προηγουμένως. Διότι οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν λιγότερες θέσεις εργασίας, είναι πιο ευάλωτες ε, στις επιπτώσεις της κρίσης δυσχερέστερα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και στον ε, παγκόσμιο ανταγωνισμό τα πάνε χειρότερα. Ποιοι είναι... Ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι ατμομηχανές της ανάπτυξης. Δείτε την Κίνα, τη Γερμανία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι. Ποιες επιχειρήσεις κάνουν επενδύσεις ε, μεγάλης κλίμακας για την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι μικρές επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου, όχι πλέον. Και τέλος, Πώ θα μπορέσει να κάνει περισσότερα η Ευρώπη για την έρευνα και την ανάπτυξη. Βεβαίως, ε, στρατηγική 2020-2050, ωραίε μεγαλοστομίε. Αλλά υπάρχουν εκθέσεις που καταδεικνύουν ότι από πλευράς επενδύσεων στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας πρώτη είναι η Κίνα, δεύτερη η Γερμανία και τρίτον οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τέλος, εάν δεν κάτσουμε κάτω μαζί να εκπονήσουμε μια στρατηγική βελτίωση της βιομηχανικής και κατασκευαστικής βάσης της Ευρώπης, με τη βοήθεια των κρατικών ενισχύσεων και της πολιτικής συνοχής, θα συνεχίσουμε να εκπονούμε θαυμάσια διανοητικώς ενδιαφέροντα κείμενα και το 2020 θα διαπιστώσουμε ότι η στρατηγική μας έχει αποτύχει. Ο Γιάννη Όλμπριχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συντονιστή που μίλησε για τον ρόλο το δικό μας, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να μην έχω πολλές γνώσεις, βλέπω όμως μια πολύ σημαντική διαφορά ε, η θέση της Επιτροπής για την μακροοικονομική ανάλυση ε, και είναι αντικειμενική γνώση αυτό ελπίζω μας λέει λοιπόν τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό για την εσωτερική αγορά και γι' αυτό υπάρχουν ε, διαβουλεύσεις, δημοσιεύσεις και κατά κάποιον τρόπο είναι η βίβλος των κρατικών ενισχύσεων για τα επόμενα 7 χρόνια. Το άλλο σκέλος είναι η πολιτική συζήτηση. Τι μπορούμε να αλλάξουμε μέσα από πολιτικές αποφάσεις και γιατί ε, πρέπει να ξέρουμε τι είναι σημαντικό και ποιο είναι το κομμάτι της αντικειμενικής ανάλυσης και γνώσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι είναι δυνατό να συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών σχημάτων. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μας δίνει ορισμένους δείκτες που είναι τα νομοθετικά κείμενα και τι θέλει από μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δείκτες, πρέπει οι πολιτικοί να τους ανακαλύψουν τους δείκτες, τι είναι αντικειμενική γνώση γνώση πράγματι. Πρέπει λοιπόν, έχουμε ορισμένα παραδείγματα, να τα κατανοήσουμε όλα αυτά. Εγώ, ε, παραδείγματος χάρη, ήμουν εισηγητής ε, και ε, πάνω σε θέματα επιχειρήσεων ε, έχουμε μία πολιτική για τις μεγάλες επιχειρήσεις από ό,τι μας λέτε που δεν είναι αποτελεσματική. Αν κατάλαβα καλά, τα, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικής ε, και άσκηση πολιτικής. Οπότε βλέπουμε πώς θα γίνει ε, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει σωστότερα τις χρηματοδοτήσεις ή αν τις δίνει σωστά οι περισσότερες επιχειρήσεις παίρνουν τα χρήματα και δεν δημιουργούν καμία θέση εργασίας και αυτό είναι σκανδαλώδες. Γιατί είναι το ότι είναι σκανδαλώδες λόγος επαρκής για να μην χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε διαφορετική λογική. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω με τη δική σας ανάλυση, να πω ότι έτσι έχει η κατάσταση. Το τι πρέπει να πράξουμε όμως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τις μεγάλες, κατά κάποιον τρόπο οι περισσότερες. Οπότε πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις γιατί συνεργάζονται με τις μικρότερες. Και αυτό χαράσει μια πολιτική και εδώ επισέρχεται η αποτελεσματικότητα και δεν είναι δυνατόν να πούμε ξαφνικά λοιπόν όχι στις μεγάλες επιχειρήσεις διότι εμείς ως πολιτικοί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Συμφωνούμε με την ανάλυση σας αλλά πρέπει να το συζητήσουμε μέσα στα πλαίσια του τριλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν φέρουμε δύο διαφορετικά κείμενα μέσα στον τρίλογο, αν ας πούμε έχουμε μία αντίθεση, ποιο κείμενο υπερισχύει, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί έτσι μπορεί να ανοίξουμε μια πόρτα, να ε, χαρούμε γιατί ε, ήρθαμε σε διαβούλευση και μετά να την ξανακλείσουμε την πόρτα. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαπραγμάτευση. Πρέπει κατά κάποιον τρόπο να λύσουμε αυτό το θέμα το ταχύτερο δυνατό. Δηλαδή να μην ε, ο τελικός αποδέκτης χάσει το το διακύβευμα. Εδώ ε, έχουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να ε, δράσουν. Ορισμένες είναι αποτελεσματικές και ξέρουμε ότι ορισμένες δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές και χρειάζονται συνεργασίες. Πώς εμείς θα δώσουμε λοιπόν ε, ενισχύσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ένα σήμα για το μέλλον ως προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να είναι κάπως πιο ευέλικτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα σύστημα ε, κρατικών ενισχύσεων ε, που να επιτρέπει τη συνεργασία των δημόσιων φορέων με ιδιωτικού φορείς και είναι δυνατόν να αλλάξουμε στάση γιατί υπάρχει, υπήρχε μια στάση που έλεγε ότι το δημόσιο ήταν καλό και το ιδιωτικό δεν ήταν καθόλου θετικό. Τώρα ε, αυτό ανατράπηκε. Αλλά τελικά τι θα πούμε. Ε, εμείς ε, θέλουμε να προάγουμε τις κατοικίες. Θέλουμε να... προάγουμε αυτή την πολιτική και ε, να υπάρχει ένας ε, συντονισμός μεταξύ των γενικών διευθύνσεων, ένας καλύτερος συντονισμός και όταν εμείς αποφασίζουμε κάτι θα πρέπει εσείς να μας ακολουθείτε. Αυτό είναι το σωστό. Ε, για αυτόν τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων θα πάρω ένα μία ακόμα ερώτηση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Όλμπριχτ. Βεβαίως, βεβαίως είναι θέμα τη Επιτροπή μα αυτό που μα απασχολεί ιδιαίτερα. Συγκεκριμένε ερωτήσει. Υπάρχουν ορισμένε περιοχέ στη Γερμανία, την Αυστρία αλλά και στην Ιταλία που στο μέλλον από εθνική άποψη βεβαίω πάνε καλά, αλλά στο μέλλον δεν θα μπορούν να λαμβάνουν όμω επιδοτήσει. Όμως αυτές οι περιφέρειες έχουν την ε, ε, το συγκεκριμένο πρόβλημα ότι συνορεύουν με, χώρες, με περιοχές σε άλλες χώρες που λαμβάνουν πολλές επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν να μεταναστεύσουν κάποια χιλιόμετρα, να περάσουν από την άλλη μεριά των συνόρων για να μπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις. Συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για την εξή πρόταση. Να υπάρχει για ορισμένες τέτοιες περιφέρειες ένα ανώτερο όριο χρηματοδοτήσεων για να μην υπάρχουν τέτοιου προβλήματα μετακίνησης από τη μία ε, πλευρά των συνόρων στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κέρστιν που ήσουν τόσο σύντομη. Να κάνω τώρα και εγώ μια ερώτηση. Πώς καθορίζει την πυκνότητα και τα όρια πληθυσμού η Κομισιόν για τις διάφορες χώρες. Και μετά ε, να δούμε. Θέλετε να απαντήσετε τώρα ή σε όλους μαζί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και για τα σχόλια που κάνατε για το πώς θέλετε να εξελιχθεί η πολιτική της Κομισιόν. Να αναφερθώ σε μερικά σημεία στα οποία αναφέρθηκαν διάφοροι ομιλητέ και που είναι νομίζω ζωτικής σημασία. Πολλοί θέσατε το θέμα των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις καθευτήρε γραμμέ για να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν δύο είδη μετεγκαταστάσεων, στο εσωτερικό της Ένωσης και εκτός Ένωσης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν θα περιέχουν μια σημαντική καινοτομία. Θα θέσουμε νέες προϋποθέσεις για τις μετεκαταστάσεις στην Ευρώπη που να είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθούν. Δεν θα επιτρέπεται μετεκατάσταση από φτωχότερη περιοχή και αν η μετεκατάσταση χρηματοδοτείται από επιδοτήσεις τότε θα πρέπει να την εξετάσουμε και να την εγκρίνουμε. Αυτό απαντά σε ερωτήσεις που έθεσαν διάφοροι και από την Επιτροπή Περιφερειών. Για τις μετεκαταστάσεις έναντι του εξωτερικού είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε αλλά η προσέγγιση μας σε αυτές τις νέες καθυντήριες γραμμές θα εξετάζει το επιπλέον κόστος για μια επιχείρηση. Εάν μια επιχείρηση μπορεί να μας αποδείξει ότι βγαίνοντας από την Ένωση θα λάβει κάποιες περαιτέρω ενισχύσεις και ότι θα είναι μεγαλύτερο το κόστος λειτουργίας της εντός Ένωσης θα επιτρέπεται. Αυτές είναι σημαντικές καινοτομίες λοιπόν που θα εισαγάγουμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις τώρα. Δεν θα επαναλάβω ήδη όσα, είπα, όσα ήδη είπα, αλλά τρία σημεία θέλω να τονίσω. Πρώτον, δεν απαγορεύεται η ενίσχυση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το τονίζω. Πρόκειται για απόλυτη παρανόηση ή παρερμηνία των προτασιών μας. Απαγορεύουμε επιδοτήσεις για αρχικές επενδύσεις στις λεγόμενες περιοχές C, αλλά υπάρχουν πολλές ακόμη δυνατότητες, ιδίως σε περιφέρειες που το Κοινοβούλιο θεωρεί πολύ σημαντικές, όπου θα μπορούν να λαμβάνουν υπό άλλες κατευθύντες γραμμές ενισχύσεις ή μεγάλες επιχειρήσεις. Περιοχές τύπου C, Γ. Είναι περιοχές που είναι λίγο πιο προηγμένες. Εκφράσατε την ανησυχία σας ότι θα απαγορεύονταν οι ενισχύσεις, οι περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις που δεν έχουν ε, περιβαλλοντικό ή στόχο ενίσχυση τη έρευνα και ανάπτυξη. Όχι. Δεν προτείνουμε εμείς ε, κατάργηση για αυτών των περιφερειών στις περιοχές α, τις φτωχότερε, όπου το ΑΕΠ είναι κάτω από το 95% του κοινωνικού όρου. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Αλλά και περαιτέρω, και αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω, εξετάζουμε δυνατότητε. ούτω ώστε υπορισμένε συνθήκε όπου κάποιε σηματοδοτήσει θα δεσμεύονται για συγκεκριμένους στόχους, να επιτρέπουμε εξαιρέσεις ακόμη και στις περιοχές αυτές τύπου C. Η πολιτική διαδικασία για την οποία μιλήσατε, όπου θα υπάρξουν νομοθετικές αποφάσεις, βεβαίως σχετίζονται με αυτήν μας την προσπάθεια. Είμαστε λοιπόν πολύ πιο κοντά ο ένας στον άλλον από ό,τι ορισμένοι μπορεί να θεωρούν και δεν έχουμε κλείσει την εξέταση του τομέα αυτού, όπως τόνισε και ο Επίτροπός μας. Τώρα, κατά πόσον ε, η κατηγοριοποίηση των περιφερειών ε, είναι συμβατές με άλλου τύπου κατηγοριοποίησης, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως, οι στόχοι είναι κάπως διαφορετικοί και γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες. Τώρα δύο συγκεκριμένα. Ορισμένοι είπατε ότι σε αυτούς τους στόχους μας, για τις κρατικές, στους χάρτες μας για τις κρατικές επιδοτήσεις, ε, να ορίσουμε ιδιαίτερο τις λεγόμενες αυτές μεταβατικές περιοχές, οι περιοχές μετάβασης. Δεν συμφωνούμε. Αν το κάνουμε αυτό, αφαιρούμε κάθε ευληγησία από τα κράτη-μέλη. Ενώ στόχος μας είναι τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα εντός κάποιου ορίου πληθυσμού να ορίζουν οι ίδιες τις περιοχές C και άρα θα μπορούν να ορίσουν εκείνες αυτές τις περιοχές μετάβασης. Θα ήταν λάθος λοιπόν να το κάνουμε εμεί αυτό, διότι κάτω από κάποιο λογικό ε, όριο πληθυσμού που είναι το 45% όπως είπαμε θα τους αφαιρούσαμε κάθε δυνατότητα ευληγησίας και το ίδιο ισχύει και για τις λεγόμενες ε, συνοριακές περιοχές και θέλω να καθησυχάσω την κυρία Βέστφαλ διότι τονίζω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν τα ίδια αυτές τις ε, συνοριακές περιοχές. Έχουν ευρεία δυνατότητα να το κάνουν γιατί είναι λίγες περιοχές που δημιουργούν πρόβλημα. Δεύτερο, εάν τις καθορίσουν έτσι, αυτές τις συνοριακές περιοχές και είναι κυρίως ε, αρκετά ευημερούσες περιφέρειες που συνορεύουν με λιγότερο ευημερούσες, αυτές οι περιοχές θα καθορίζονται με κάπως λιγότερο γενναιόδορο τρόπο από ό,τι σήμερα, αλλά θα συνεχίσουν να καθορίζονται. Είναι λοιπόν θέμα επικουρικότητας πιστεύω. Η Κομισιόν να κάνει μόνη της τον πλήρη καθορισμό των περιχών αυτών, αφαιρώντας κάθε δυνατότητα από τα κράτη-μέλη να παρέμβουν στον τομέα αυτό. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερα λοιπόν τα κράτη-μέλη να έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά στα πλαίσια γενναιόδωρων κανόνων. Επιλέξαμε αυτή τη δεύτερη λύση. Τώρα δεν είναι δικό μου θέμα να σχολιάσω τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Κοινοβούλιο, αλλά τονίζω ότι και μετά αυτή τη συζήτηση βεβαίως είμαστε ανοιχτοί για τη συνέχιση του διαλόγου, για ασθενή συνεργασία και με τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Regio, αλλά και με εσά. Έγιναν διάφορες ερωτήσει για άλλα μέσα ενίσχυση για την ε, πληροφορική, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Βεβαίως έχουμε παρόμοιο διάλογο και για τα θέματα αυτά για να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των πολιτικών και η κυρία Χούμπνερ με ρώτησε από πού προκύπτει αυτό το κατόφλιο πληθυσμού. Είπα ότι θα εναρμονίσουμε την πολιτική μας με την ισχύουσα πολιτική για τα κατόφλια πληθυσμών που είναι κάτω λοιπόν από το 50% προσπαθούμε να εξορροπήσουμε την ε, αποτελεσματική χρήση πόρων έναντι της ευρύτερης ε, χορήγησης πόρων και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτές μας τις προσεγγίσεις, διότι με αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη θα έχουν ε, ευρύτερη δυνατότητα να καθορίσουν την περιφερειακή τους πολιτική. Έχουν μειωθεί οι ανισότητες στην Ευρώπη, έχουμε πολύ λιγότερες πολύ φτυχές περιοχές από, πολύ φτωχές περιοχές από ό,τι πριν από μία δεκαπενταετία. Έτσι λοιπόν, εφόσον το συνολικό ποσό είναι σταθερό, τα κράτη-μέλη θα έχουν ευρύτερη δυνατότητα να ενισχύσουν διάφορες ε, περιφέρειες στα πλαίσια της ε, ε, πολιτικής συνοχής της Ένωσης. Η κυρία Χιούμπνερ. Για το θέμα του ποιο είναι πιο σημαντικό στο Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή θα πρέπει να επανέλθουμε. Νομίζω ότι θα ήθελα και εγώ τώρα να ε, σχολιάσω μερικά σημεία. Ε, καταρχήν το θέμα δεν είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι κακές όπως είπατε καθόλου. Καθόλου μάλιστα το θέμα του στόχου της πολιτικής συνοχής μας απασχολεί και επίσης το ότι έχουμε ένα καθορισμένο όγκο ε, πόρων το που δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε ε, χωρίς να θεσπίσουμε ορισμένα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε και στον τρίλογο. Πρέπει να δράσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και κανείς δεν θέλει απόλυτα ανοιχτή διαδικασία σε αυτό το τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Η πολιτική συνοχής πρέπει να είναι μια πολιτική που να παροτρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη μέσα σε, στην περιφέρεια. Ε, είναι ωστόσο αναπόφευκτο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πίεσης που προκύπτουν από το ε, πακέτο ε, το οποίο πρέπει να προγραμματιστεί για να προχωρήσουμε ε, προς μια εξέλιξη. Επίσης ε, πρέπει να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων παράλληλα, ακριβώ παράλληλα, γιατί καθορίζονται οι κανόνες της κρατικής ε, ενίσχυσης σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της περιφερειακής πολιτικής και μετά χρησιμοποιείται η διαδικασία της έγκρισης των χαρτών ε, κατά κράτος και αυτό πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στο τέλος να υπάρξει ένα σωστός προγραμματισμός. Ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε έναν συντονισμό ε, των ε, όσων θα ε, πρόκειται να λάβουν επιδοτήσεις για να έχουμε μια πολιτική συνοχή στην οποία θα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεσμικό όργανο να ε, μπορέσει να αποφύγει τις διάφορες ανομαλίες και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να πράξουμε. Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι περιοχές ενδεχομένου κινδύνου και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό στις περιφέρειες και να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά όσο θεσπίζουμε τη διαδικασία διαδικασία ε, της, ε, του καθορισμού των κατευθυντηρίων γραμμών. Να εκπονήσουμε λοιπόν την τελική θέση ε, για, τις, για τον καθορισμό των look για την ε, διαδικασία των ε, ελέγχων που πρέπει να γίνουν σε διάφορες ζώνες που πρέπει να εξετάσουμε την τελική, ε, τον τελικό καθορισμό των χαρτών. είναι ευθύνη μας να το πράξουμε αυτό για να δούμε ποιο θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα γιατί θα πρέπει να μην υπάρχουν οι ανομαλίες τις οποίες θέλουμε να αποφύγουμε. Κύριε Ντερανό, σε ευχαριστώ που λαμβάνω και πάλι το λόγο. Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό το αν γίνεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή για νέα παραγωγή όπως τις ε, ανθρακούχες ίνες ε, που θα μπορούσε να είναι και το υλικό του μέλλοντος. Αν δεν μπορούμε εδώ στην Ευρώπη να μπορέσουμε να το παράγουμε, τότε οι Κινέζοι οι Αμερικανοί θα το κάνουν. Θα πρέπει αυτά να τα καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε και απευθύνομαι στην Επιτροπή. Για αυτό το θέμα ακριβώ οπωσδήποτε οι μεγάλες εταιρείες μας θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα αυτό γιατί δεν μπορούν να το κάνουν από μόνο οι μικρές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο και το είπαν και αρκετοί που πήραν τον λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συνδεμένες συχνά με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν για να δημιουργηθεί αυτή η σύγκληση ανάμεσα στις μικρές μεγάλες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό παρακαλώ προσέξτε για το μέλλον των βιομηχανικών της Ευρώπης. Αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία. Εκεί δίνουμε τη μάχη μας ώστε να μπορέσουν οι μεγάλες επιχείρησεις να επιλεχθούν. Εντάξει κάτω από όλες τις συνθήκες βέβαια. Όχι να επιλέξουμε για όλα τα θέματα, για κάθε θέμα όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να στηριχθούμε σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης. Κάτι ακόμα για τις ε, περιοχές ε, γάμα ε, ε, και αυτές υποφέρουν. Είναι αγροτικές πολλές φορές ε, περιοχές που έχουν είτε είναι οποιοδήποτε θέμα μπαίνει στη μέση συνδρομικό, οδικό κλπ. Αντιμετωπίζουν διπλές δυσκολίες. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές με τις ίδιες με τρόπο όπως και με τις περιοχές της Α γιατί είναι ανάμεσα στο 75% και στο 80% στο μέσο ΑΕΠ της Ευρώπης. Έτσι. Επειδή ε, ήδη έχουμε πάρει από το χρόνο ε, ψηφοφορία, παρακαλώ να είστε σύντομοι και να μην επαναλάβετε θέματα που έχουν ήδη αναφερθεί ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για τον συνδυασμό της περιφερειακής και ανταγωνιστικής πολιτικής, πολιτικής ανταγωνισμού. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Όλμπριχτ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, σωσμένες ε, περιφέρειες Όπω στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει μόνο μία ή δύο μεγάλε επιχειρήσει. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτέ τι μεγάλε επιχειρήσει για να πάρουν μαζί του και τι μικρομεσαίε. Και θα ήθελα να μου πείτε τι θα γίνει ε, με τι λεγόμενε περιοχέ Α. Πώ θα ληφθούν υπόψη του μεταβατικού κανονισμού. Ευχαριστώ. Η Μόνικα Σμόλκοβα. Σας ευχαριστώ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 Euh, Ευχαριστώ να υποστηρίξω την πρόταση του συναδελφού του ε, για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να είμαστε και παρόντες στην συζήτηση αυτή. Πολύ σημαντικό είναι όλα αυτά να συνδυαστούν, δηλαδή η πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανταγωνισμό, για τι περιφέρειε. Είναι διάφοροι πυλώνε μια πολιτική, για να δούμε πόση βοήθεια, πόση συγχρηματοδότηση και για τι περιφέρειε αυτέ που επιτρέπονται ακριβώ να διονται από τα κράτη μελη έτσι, να υπάρχει μια συνοχή. Και βλέπω ότι η αυτή θρηματίζεται και δεν λαμβάνει υπόψη αυτές οι διάμεσες περιοχές και η πολιτική συνοχή που προτείνει η Επιτροπή ακριβώς το 2014-2020. Χρειάζεται να συνδυαστούν όλα αυτά, να συγκλίνουν και ακόμα κάτι το δεύτερο, μια σύγκληση είναι με τις συνθήκες. Τι κάνουμε ακριβώς με τις συνθήκες συνθήκη της Αβώνας και με τις μειονεκτικές και να δούμε και τις νησιωτικές περιοχές που χρειάζεται και πάλι να αναδυθούν σε σχέση με τις υπόλοιπες με πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και να είναι ίσες αυτές τις περιοχές απέναντι σε οικονομικά θέματα και οικονομικές δραστηριότητες όταν είναι μικρά νησιά ακριβώ που καταλαβαίνουμε τον ευαίσθητο τους χαρακτήρα όσον αφορά αυτό το, την οικονομική πτυχή. Χρειάζεται λοιπόν μια σύγκληση ανάμεσα σε αυτά δύο και οπωσδήποτε είμαστε δίπλα στην Επιτροπή, θα μπορείτε να συναντιέστε και θα μπορούσατε να έχετε και μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή. Merci. Ο πάμενος ομιλητής, ε, σας ευχαριστώ. Θα πρέπει σιγά σιγά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διάφορες ρυθμίσεις και νομικές και του μάλλον και του προπολογισμού, μάλλον αυτά γίνονται, αλλά αυτά που δυναμώνουν την περιφερειακή πολιτική και πρόκειται για ένα ακόμα στοιχείο πάντως που θα μπορούσαμε να κάνουμε το αντίθετο για να εξηγιάνουμε αυτή την πολιτική. Θα πρέπει να προσέξουμε αυτές τις αρχές που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Αλλά οτιδήποτε και αν υποστηρίζει κανείς βλέπουμε ότι μειώνεται και ο όγκος και η ποσότητα ακριβώ των ενισχύσεων. Και ο πρόεδρος ε, των περιφερειακών κύριος Διδιέ ας ε, μας τα είπε αυτά μα είπε ότι ε, αυτή η ιδιαίτερη μείωση και στις πιο ευάλωτες περιοχές θα πρέπει να αντισταθούμε κυρίως σε παρόμοια εποχή κρίσης και πρόκειται για μια πρόταση που δεν στέκει εδώ σε σχέση τουλάχιστον με τις ανάγκες. Αντίθετα θα έπρεπε να ενισχύσουμε αυτές τις ενισχύσεις να πετύχουμε τους στόχους και που τους υπενθύμησε ο εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειών και Α, απαλού όμως βλέπουμε ότι έγινε εντελώς το αντίθετο. Είναι θέματα που δημιουργούν προβλήματα στην πρόταση αυτή. Αναφέρθηκε γιατί υπάρχει μια κάποια ανισότητα σε διάφορες πτυχές ανάμεσα στις κατηγορίες περιφερειών και μέσα και στην αυτή κατηγορία περιφερειών τι προβλεπόταν, σας λέω σαν παράδειγμα, ότι όσοι φεύγουν ακριβώς από την ε, στόχο σύγκλησης, ε, τι γίνεται, ότι είναι θετικά τα πράγματα, αλλά εκείνες που είναι μέσα εκεί, αντίθετα, βλέπουμε ότι θα επιβαρυνόταν και κάτι τέτοιο δεν μπορούμε που δεν είναι να το δεχτούμε. Σχετικά με τις μεταγκαταστάσεις, ε, σίγουρα αυτά τα μέτρα θα ενισχύσουν τις μετακαταστάσεις και γι' αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί μια κάποια ρύθμιση που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις εκείνες που μεταγκαθίστανται και μάλιστα τουλάχιστον για πέντε χρόνια τουλάχιστον που θα έχουν πάρει ενισχύσεις και να του ζητείτε και να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα που έχουν λάβει και για τις περιφερειακές περιοχές. Αυτό το ερώτημα το υποβάλλω στην Επιτροπή. Τι προβλέπετε σχετικά με αυτό το μπόνους που δινόταν στις εν λόγω περιοχές. Διατηρείται αυτό, ισχύει, είτε μειώνεται κατά το ίμιση, όπως ε, έχω νομίζω ότι συμβαίνει. Αυτές οι ερωτήσεις θα ήθελα να υποβάλλω όσον αφορά το θέμα και νομίζω ότι θα πούμε κι άλλα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των μεγάλων επιχειρήσεων. Από ό,τι είδα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, φαίνεται ότι η τάση είναι προς ε, ε, την ενίσχυση των μεγάλων εταιριών. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες εποφελούνται ωστόσο από τις μεγάλες ορισμένες περιοχές γιατί είναι μέλος της αλυσίδας παροχής. Οι μεγάλες ε, εταιρείε έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις περιφέρειες γιατί ε, αναπτύσσουν, βοηθούν την ανάπτυξη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, στο, στην βόρεια, βορειοανατολική Ουαλία υπήρχε μία, ένα μεγάλο κλαμπ το οποίο ήθελε να ε, χρησιμοποιήσει τις ε, μεγάλες εταιρείες για να ενισχύσει, για να μπορέσει να αναπτυχθεί οικονομικά και έτσι ενισχύεται η τοπική οικονομία. Δεν είναι μόνο θέμα ιδιωτικού τομέα και ανάπτυξής του, αλλά είναι θέμα χρησιμοποίηση σωστή των προτάσεων και οι προτάσεις έρχονται κατευθείαν στις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν ολόκληρη την περιφέρεια, ολόκληρη τη ζώνη της περιφέρειας η οποία θα αναπτυχθεί με τη σειρά της και αυτός είναι ο ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ορισμένε στοχευμένε εξαιρέσει, Γιατί έγινε ήδη λόγο γι' αυτό. Ε, είναι κάτι το οποίο το σκεφτόσαστε ήδη και θα έχετε κάποιε ιδέε και προτάσει για τι στοχευμένε αυτές εξαιρεσει. Σω θα μπορούσατε να μας ε, μιλήσετε περαιτέρω για αυτή την πρόταση. Οι κρατικές ενισχύσει για τι περιφέρειες είναι ένα από τα κύρια όργανα για την επίτευξη της συνοχής ε, τη οικονομική στην περιφέρεια και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία και να έχει μια συνεκτικότητα. Βέβαια οι συνθήκες πρέπει να είναι τώρα πολύ πιο αυστηρέ και χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και νομίζω ότι ο συντονισμός των κρατικών ενισχύσεων με άλλες πολιτικές, όπως είπαν πολύ προλαλήσαντες, είναι κάτι το σωστό. Ε, θα ήθελα να μιλήσω ε, για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που συχνά ε, θα μπορούν να γνωρίσουν φραγμούς σημαντικούς. Ας μην το κάνουμε αυτό, διότι είναι καλύτερα να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα ενγέρος και όχι όταν θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις σχετικά. Δεν χρειάζονται περισσότερα, ε, περισσότερες ε, διοικητικές απαγορεύσεις. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ε, παροτρύνουμε, να εξηγούμε, να δείχνουμε ότι αυτά που συμβαίνουν είναι ε, για την ανάπτυξη της περιοχής, γιατί δεν μπορούν να παρασχεθούν τα κλασικού τύπου δάνεια, παραδείγματος χάρη, ή να χρησιμοποιηθούν οι βοήθειες όπως παλιότερα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι φορτίο, είναι βάρος και για τις κυβερνήσεις, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν απαραίτητο, πιστεύω, να υπάρχουν αυστηρές συνθήκες, οι οποίες να θεσπιστούν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για δημόσιες ενισχύσεις. Ε, ακριβώς είμαστε υπέρ των πολιτών ε, της πλειονότητας των πολιτών. Ε, θα μιλήσω για τη Μαδρίτη με περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους η περιοχή που αυτή τη στιγμή όμως αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη ανεργία και ταυτόχρονα από τις περιφέρειες όπου υπάρχουν δυνατότητες όσον αφορά την κοινοτομία, αλλά δεν έρχεται η ενίσχυση. Θα ήθελα τον κύριο Μάρτιν βάσει του άρθρου 107.3 της συνθήκης της ιδρυτικής πράξης ακριβώς ε, υπάρχουν και άλλοι δείκτες εκτός από το ΑΕΠ που αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα. Να μπορέσουν αυτές οι ενισχύσει να φτάσουν σε περιοχές όπως η Μαδρίτη. Ναι, ολοκληρώσαμε τον κατάλογο. Παρακαλώ την Επιτροπή να απαντήσει όπως επίσης και την Επιτροπή να κάνει ένα σχόλιο. Ποιος θα αρχίσει? Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Δεν είναι δυνατό καθόλου να απαντηθούν όλες, αλλά θα σας απαντήσω στα πιο σημαντικά θέματα, ελπίζω. Και ίσως πρέπει να πω ότι βεβαίως λαμβάνουμε πλήρως υπόψη των στόχων της περιφερειακής πολιτικής και πράττοντας το λαμβάνουμε υπόψη και τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και όχι περισσότερη ε, περιορισμοί αλλά οπωσδήποτε δεν θέλουμε να, να παραβλάψουμε ούτε την περιφερειακή πολιτική ούτε την πολιτική ανταγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει υπόψη του τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αλλά πρέπει και εμείς να λάβουμε υπόψη τις ε, ε δαπάνες. Δεν είναι ταυτόσιμα ε, τα, τα δεν είναι ταυτόσιμη στόχη ορισμένων κρατών που θέλουν να έχουν τις περισσότερες δυνατές επιδοτήσεις. Πρέπει να δούμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν μεγάλη δυνατότητα ε, δαπανών ενώ άλλα έχουν πάρα πολύ μικρή ε, τέτοια δυνατότητα και εμείς πρέπει να είμαστε συνετοί και να προσέχουμε το πώς θα γίνουν οι επιδοτήσεις. Ε, υπάρχουν μπροστά μας πολλά χρόνια ύφεσης και πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε τους σπόρους μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεσπίσουμε κριτήρια για τις χώρες εκείνες που έχουν μικρή ε, δυνατότητα. Ε, είναι πιο φτωχές χώρες. Δεν πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα κατά των φτωχοτέρων χωρών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νέες πραγματικότητες της Ευρώπης που δυστυχώς τις αντιμετωπίζουμε όλοι από κοινού. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε, ορισμένες, σε συγκεκριμένες περιφέρειες και γι' αυτό λαμβάνουμε ορισμένα μέτρα τα οποία ξεπερνούν τα, ή αλλάζουν τα σημερινά μέτρα ε, θεσπίζοντας ορισμένες, ορισμένους κανόνες ε, ε, γιατί υπάρχουν ε, παραδείγματος χάρη ε, περιφερειακές περιφέρειες και περιφέρειες στην υπηρετική Ευρώπη και είναι εντελώς διαφορετικός ο συσχετισμός μεταξύ των θα πρέπει τώρα να αναφερθώ στο, στην ανάγκη διαφάνειας την οποία ανάφερε ένας συνάδελφος. Ε, εμείς προτείναμε και θα επιμείνουμε από αυτού σαν γενικό κανόνα όχι μόνο για τις κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακής πολιτικής αλλά για όλες τις κατευθυντήριες γραμμές να έχουμε τη σωστή εικόνα του αποδέκτη γιατί είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να δουλέψει το σύστημα ε, πολλές φορές ε, μπορείτε να δοκιμάσετε έκπληξη γιατί ήδη δεν τα γνωρίζουμε όλα τώρα στην υπάρχουσα φάση των κανόνων. Όμως ε, θα προχωρήσουμε τον έλεγχο και θα έχουμε μια καλύτερη τοποθέτηση ως προς αυτό το θέμα. Ο Νίκος μίλησε για το, τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι συνομοθετική διαδικασία ε, για την περιφερειακή πολιτική αλλά και για άλλες ε, πολιτικές. Πρέπει να δούμε ότι και να, να σας ε, ε, εξηγήσουμε το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη θέσπιση της πολιτικής του ανταγωνισμού ε, ασχολούνται με όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε και έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις με συναδέλφους σε άλλα θεσμικά όργανα για να εδρεώσουμε τη θέση μας επί των ε, κανόνων που δημιουργούμε και θέλουμε να έχουμε από τη μία πλευρά μια ευρύτερη πολιτική σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο ανταγωνισμού. Ε, νομίζω ότι παραδεχόμαστε οπωσδήποτε ότι είναι δύσκολο να συμφιλιώσουμε αυτές τις δύο τάσεις αλλά θέλουμε τουλάχιστον να ισοθήσουμε να εξελιχθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν ορισμένοι συνομιλητές σε αυτήν την ε, συζήτηση που έχουμε που έχουν διαφορετικούς στόχους. Δεν προάγουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την εσωτερική αγορά και την εξέλιξή της ούτε την πολιτική συνοχή καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θέλω να επανέλθω. Ε, το θέμα των δικτών ε, και του ΑΕΠ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα ουσίας γιατί η κατηγοριοποίηση των περιοχών για την πολιτική συνοχή βασίζεται στο ΑΕΠ και βεβαίως ε, έτσι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν ανισομέρειες με τον στον τρόπο που χαρακτηρίζουμε τις περιφέρειες ότι χρησιμοποιούμε τους ίδιους δείκτες και δεν γίνονται διακρίσεις. Είναι μία από τις τις ε, θέσεις κλειδιά που έχουμε για το χαρακτηρισμό των κατηγοριών ε, για τις κατηγορίες των περιοχών και ε, πρέπει να πω ότι είδαμε στις συζητήσεις για την πολιτική συνοχής ότι έχουμε ορισμένα αποτελέσματα των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβολίου και ε, έχουμε ορισμένες ε, σύμφωνα με αυτά διαφοροποιήσεις τύπων περιφερειών ε, παραδείγματος χάρη υπήρχαν πρώην ε, συγκλήσεις οι οποίες ε, στην μεταβατική κατηγορία θα χρησιμοποιηθούν και υπήρχαν επίσης για την επόμενη περίοδο μεγαλύτερες περιφέρειες οι οποίες θα επισέλθουν στην ίδια κατηγορία. Ε, για να υπάρχουν επίσης περιφέρειες του phasing out και θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε κατηγορίες συγχρηματοδότησης ε, ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις που θα θεσπίσουμε. Είναι πάρα πολύ σύνθετη αυτή η διαφοροποίηση και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πλήρως τις αντιστοιχίες που θα υπάρχουν με την παροχή ενισχύσεων ε, στην κάθε περιοχή. Ανάλογα με τις επιλογές που θα πράξουμε δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο και ε, υπάρχει και το θέμα των περιφερειών που έχουν ε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τα δούμε σαν ε, μειονεκτήματα ε, και υπάρχει μια ειδική μεταχείριση για ορισμένες περιφέρειες ε, ειδικά χαρακτηριστικά τα νησιά οι ορεινές περιοχές οι απομακρυσμένες περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και εκεί υπάρχει μια ευελιξία για τον καθορισμό των ποσοστών συγχρηματοδότησης που πρέπει να θεσπίσουμε. Χρειάζεται ένας προκαθορισμός του ποια θα είναι η μεταχείριση της περιφερειακής ενίσχυσης σε αυτό το επίπεδο. Και τελικά ένα τελευταίο σημείο που αντιστοιχεί ε, στα όσα είπε ο κύριος Μπον. Είπατε ότι πρέπει να εξετάσουμε το όλο πλαίσιο, δηλαδή να δούμε τι, ποιος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό το συζητήσαμε στον Τρίλογο. Είναι πολύ σημαντικό να χαρακτηριστεί σωστά η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες. Ε, και υπάρχουν ορισμένες προτεραιότητες ε, στον καθορισμό των ε, κατευθυντηρίων γραμμών που θα καθορίσουν τελικά το καθεστώς που θα διέπει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα έπρεπε να μπούμε στα πλαίσια αυτής της κρίσης, να την καταλάβουμε αυτή που περνάει η Ευρώπη. Και χρειάζονται και δημόσιες παρεμβάσεις. Όχι, δεν είναι εκείνες που θα αναθερμάνουν την αγορά και μας λείβει ιδιαίτερα το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 2014-2020. Το Πακίνοβούλιο ελπίζω να μπορέσει να πει και τη δικιά του την άποψη και έτσι η δημόσια παρέμβαση που συμπληρώνει εκείνη των κρατών είναι αποτελεσματικότερη γιατί αποτελεί ε, κάτι το πολύ σημαντικό σαν ενέργεια για το μέλλον των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δεύτερο, για τη συνοχή τώρα ανάμεσα στις διάφορες κατευθυντές γραμμές και τα ε, διαχωτικά ευρωπαϊκά ταμεία που είναι υπέρ της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σίγουρα χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα όμως ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης για να μπορέσουν ε, να αναπτυχθούν μια λογική συνοχή ανάμεσα στα δύο συστήματα και να επιμείνω όσον αφορά τον αγροτικό χαρακτήρα της Ευρώπης, έτσι το Ρουράκτ ε, με 50 περιφέρειες ευρωπαϊκές ε, και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εξόδου και είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις αστική, αστικές περιοχές και αγροτικές γιατί χρειάζεται ενίσχυση εκεί στις αγροτικές περιοχές να διατηρηθούν εκεί οι πληθυσμοί να υπάρξει ισορροπία, να διατηρηθεί ισορροπία. Αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω μετά από την όλη συζήτηση αλλά παρακαλώ από την Επιτροπή τους παρισταμένους είδατε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να επιλέξουμε τις κατάλληλες εταιρείε. Θα πρέπει να καταλάβουμε αυτή την κατάσταση που έχει ένα ειδικό χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Και βεβαίως εκφράζω την ευχή ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να συνεχιστεί. Η Επιτροπή και ιδιαίτερα ο κύριος Κόπμαν δήλωσε τη διαθεσιμότητα περαιτέρω ανταλλαγής απόψεων. Θα υπάρξει προφορική ερώτηση για την Ολομέλεια. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε και θα ολοκληρώσετε τέλη Μαρτίου τη συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ίσως μετά μπορούμε να επανέλθουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα που προέκυψαν και από τον τριμερή διάλογό μας για το νομοθετικό πλαίσιο της επόμενης περίοδου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που δείχνετε τέτοια θετική διάθεση συνεργασίας. Καταλαβαίνουμε το ρόλο της ε, Κομισιόν για τον ανταγωνισμό. Πιστεύουμε όμως ότι αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικός για την αποτελεσματικότητα και του δικού μας τομέα. Γι' αυτό είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να ελέγξουμε αν λειτουργούν οι ηλεκτρονικές σας κάρτες ψηφοφορίας, κάνουμε λοιπόν μια εικονική ψηφοφορία, άρχεται. Είναι λίγο αργό αλλά λειτουργεί. Oh, you have already there. Okay. You knew already. Okay, it, not everybody voted. Ψηφίσατε όλοι, όχι. Από ό,τι κατάλαβα, τρία ή τέσσερα άτομα δεν θέλησαν να ψηφίσουν. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι λειτουργούν όλες οι κάρτες. Έχουμε λοιπόν την απαλλαγή. Έκθεση Όλμπριχτ. Συμβαστική ένα ποιήν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5 είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιημένη τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται οπότε έχουμε μια προφορική τροπολόγηση Τη τροπολογία 9 είναι κανείς κατά όχι ωραία ψηφίζουμε τροπολογία 9 τροποποιηθήσα υπέρ υπέρ έλεγα κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 όπου επίσης έχει τροποποιηθεί προφορικός είναι κατά κανείς προφορική τροπολόγηση, ωραία τροποποιημένη τροπολογία 10 υπέρ κατά θα πρέπει να ελέγξουμε. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ 21 κατά. Ε, συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την γνωμοδότηση. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. πέρασε 40 υπέρ ένας κατά. Περνάμε τώρα στην έκθεση Ρίκα Μάνερ. Μπορούμε να ψηφίσουμε Ρίκα. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά. Απορρίπτεται αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. 8 λέω. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται πιστεύω. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. 11 λέω. Ωραία. Να ελέγξουμε την τροπολογία 10 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Την 11 την ψηφίσαμε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 40 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 24-18 τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Υπάρχει μια προφορική τροπολόγηση της τροπολογία 5 της συμβαστική. Έχει κανεί αντίρρηση? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική 5 τροποποιηθήσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 61. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 28-14. Ορίστε. Α. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, να ελέγξουμε την 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 προς 18. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά να την ελέγξουμε. Την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 24 προς 18. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ε, συγγνώμη 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται 39 υπέρ κατά 3. Οπότε λίγη η ψηφοφορία. Τώρα έχουμε την πρώτη μας συνάντηση με τον κύριο Ραμόν Λουίς Μπαλκάρθελ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών. Δεν έχει διακοπεί η συνεδρίαση. Παρακαλώ. I like Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλωσορίζω ολόθερμα για πρώτη φορά με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών, τον Ραμόν Λουίς Βαλκάρθελ. Και τον καλό να πάρει το λόγο ευθύς αμέσως και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτή τη συμφωνία της 8 Φεβρουαρίου από τους ηγέτες ε, Κατών και κυβερνήσεων για το πολιετές πλαίσιο 2014-2020 θα μπορούσε κανένα να σκεφτεί ότι τα πάντα αναφέρθηκαν αλλά Δυστυχώς δεν πρόκειται για κάτι παρόμοιο. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσκαλούν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πετύχουν μια συμφωνία όσο γίνεται συντομότερα, όπως το τόνισε αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πραγματικές διαπραγματεύσεις τώρα ξεκινούν. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας συγχαρτήρια για δύο λόγους. Αφενός γιατί υποστηρίξατε σταθερά τις θέσεις σας για το δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο και επίσης για το πόσο προχώρησε η υπόθεση στο πλαίσιο αυτών διαπραγματεύσεων με τον τριμερή διάλογο για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μερικοί έχουν την τάση να λησμονούν ότι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 2005 και του 2006. Από τότε η συνθήκη της Σαββόνας δίδει κοινές αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τα δούμε πώς θα εγκρίνει το πολιετές πλαίσιο ακριβώς που υιοθέτησε το Συμβούλιο και επίσης μια δυνατότητα συναπόφασης του νομοθετικού ε, συνόλου σχετικό με την πολιτική συνοχής. Και τώρα είναι μια αποφαστική καμπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ακριβώς είναι το θεσμικό όργανο που μπορεί να θέσει την σφραγίδα του σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τις περιφέρειες της Ευρώπης. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Επιτροπή Περιφύριων ε, συμμετείχε στο σύνολο των συζήτησης με το πλαίσιο το Δεκέμβριο του 2011 και μια, διάφορες εκθέσεις για όλες τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις ε, μελλοντικέ πολιτικές ε, της περίοδου 2014-2020, την ΚΑΠ, την πολιτική Συνοχής και διάφορα άλλα σημεία. Και επίσης επεξεργαστήκαμε μια αναθεωρημένη έκθεση σχετικά με το πολιετές πλαίσιο αυτό. Τον Οκτώβριο το κάναμε και πριν τις 22 Νοεμβρίου πριν από τη συνάντηση του Συμβουλίου και επίσης ακόμα μια απόφαση για την πολιτική συνοχή. Και οι συγητές μας ήταν σε άμεση επαφή με τους συναδέλφους τους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι είμαστε γιατί συνεργαστήκαμε γιατί πολλές από τις συστάσεις ας πούμε για τροπολογία στα νομοθετικά πλαίσια που απαριθμίσαμε ακριβώ ε, στις εκθέσεις μας και πολλά από αυτά που μας απασχολούσαν ε, έτυχαν θετικής υποδοχής από την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή. Η συζήτηση αυτή τώρα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί το σημερινό οικονομικό πλαίσιο δεν είναι και τόσο θετικό και το λέμε ότι δυστυχώ χειροτερεύει πολύ κατάσταση σε τοπικό επίπεδο. Η πολιτική συνοχή αποτελεί ένα εργαλείο σημαντικότατο για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση επιτόπου και να πετύχουμε του στόχου μας, του οποίου έχουμε θέσει με στόχο το 2020. Όλα αυτά αυτά τα διαφορετικά κονδύλια είναι το 1 τρίτο και για τα μισά τουλάχιστον κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θέματα καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βοήθεια την κοινωνική που είναι όλα αυτά σημαντικά για τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Όλα αυτά. Γνωρίζετε πολύ από εσά ότι χωρίς διαδοτικά ταμεία επουδενή δεν θα υπήρχαν επαρκεί επενδύσει. αλλά σίγουρα θα υπήρχε κίνδυνος να λιμνάσουμε οικονομικά και σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές τα όσα υπόθηκαν εκεί θα πρέπει να δούμε τώρα πώς το θεωρούμε μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι θα σας πω γιατί η απόψή μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε μόνο κάπως λογικά, σύμφωνα με τη λογική ικανοποιημένοι με αυτά να υποστηρίξω τα θετικά της συμφωνίας στο ε, Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό. Να πω καταρχήν ότι ο προϋπολογισμός βέβαια ελαφρώς μειώθηκε σε σχέση με ε, ε, προηγούμενα 225 εκατομμύρια αφαιρέθηκε ένα σημαντικό ποσό σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η περικοπή αυτή σε σχέση με τη σημερινή περίοδο είναι 29 δισεκατομμύρια. 18% λιγότερο και οπωσδήποτε βέβαια πρόκειται για μια σημαντική μείωση, περικοπή και θα πρέπει όμως και να υπενθυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο και λιγότερο πολλά κράτη-μέλη ήταν υπέρ του να διαγραφεί εντελώ η περιφερειακή πολιτική. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αντιστάθηκε σε αυτήν την πίεση η περιφερειακή πολιτική απέναντι στους αντιπάλους, στους εχθρούς της ε, συνοχής και μαζί με την ΚΑΠ ήταν από τους κύριους πυλώνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Κάτι ακόμα να σας προσθέσω η συμφωνία για τις και προοπτικες προοπτικές 2014-2020 έτσι τουλάχιστον μπορούμε να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα και σχετικά για την, με τη σταθερότητα του πολιτού σχεδιασμού ενώ δεν είναι εύκολος στόχος να επιτευχθεί μπροστά στις αντιθέσεις πολλών από τους 27. Και ακόμη κάτι. Ανάμεσα αυτά που θα πρέπει να τονίσουμε στη συμφωνία, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και ότι είμαστε ικανοποιημένοι για τη διατήρηση της όλης αρχιτεκτονικής της περιφερειακής πολιτικής, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα για την κατηγορία των μεταβατικών, των σε μετάβαση περιοχών. Και η Επιτροπή Περιφερειών έδωσε αγώνα για να δημιουργηθεί μια κατηγορία που ακριβώς που να έχει μια αντιμετώπιση δίκαιη απέναντι σε περιοχές που οποίες έχουν ενδιάμεσο ποσοστό ανάπτυξης ανάμεσα στο 75% και στο 90% του κοινοτικού ΑΕΠ και να αποφύγουμε στρεβλώσεις σημαντικές απέναντι σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς ε, σε μάχησε μαζί μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν σημαντικότατο σύμμαχος. Και τα τρία προηγούμενα σημεία που είπα, θα σας πω ότι θα μπορούσαμε να τονίσουμε και τη νέα πρωτοβουλία της απασχόλησης των νέων για τις περιοχές που έχουν ε, τουλάχιστον 25% ε, ανεργία νέων και εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα κάθε πρωτοβουλία που είναι υπέρ της επίλυσης του προβλήματος αυτού. Και πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίναμε ένα ψήφισμα σχετικό και υποστηρίζαμε το σχέδιο της εγγύησης ε, αναζήτησης εργασίας για τους νέους και για αυτή την πρωτοβουλία. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε τοπικούς φορείς. Ε, κάτι ακόμα το σίγουρο είναι η δημιουργία του μηχανισμού του κατάλληλου για την Ευρώπη που τίνει προς χρηματοδότηση υποδομής του, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών παρόλο που 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την πρώτη επιτροπή μειώθηκε το ποσό αυτό αλλά η πολιτική αυτή σίγουρα από 12 ε, από περίπου 13 δισεκατομμύρια θα περάσει σε από 12,9 θα περάσει στα 29. Και είναι κάτι το θετικό το άνοιγμα ακριβώ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά μια ευκαμψία και ευληγησία. Η 109 παράγραφος των συμπρασμάτων λέει ακριβώς με αυτούς τους όρους ότι γίνεται περισσότερη ευληγησία. Και ήταν η νίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί επέμεινε σε αυτό το μέτρο πολλές φορές και εμείς χαιρόμαστε από την Επιτροπή Ελευθεριών με αυτή την πρόοδο γιατί έτσι ζητήσαμε και μία άμεση αναθεώρηση του πλαισίου του δημοσιομικού του πολίτους. Είναι κάτι το αναγκαίο και το δίκαιο επίσης γιατί θα πρέπει, δεν θα είναι σίγουρα η κατάσταση ίδια μέσα σε τέσσερα χρόνια και τότε θα πρέπει ορισμένες ε, ελλείψεις να τις διορθώσουμε μέσα στον προπολογισμό. Και έχω γνώση των δυσκελιών για να πετύχουμε τη συμφωνία με 27 κράτη-μέλη. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η συμφωνία του Συμβουλίου ήταν και καλύτερη και ότι δεν υπάρχουν και δυνατότητες διαπραγματεύσεων. Εδώ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, συμφωνούμε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, δύσκολες, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε μία απόρριψη της συμφωνίας, γιατί η οικονομική κρίση θα χτυπάει πάντα την πραγματικότητά μας και θα ε, είναι παραγωνοπιστό δρόμησης. και εδώ ολοκληρώνω εδώ εμείς θα θέλαμε να υπάρξουν ορισμένε διορθώσεις επιγραμμίσεις και ανέφερα το θέμα της ευληγησίας εντάξει θα μπορούσε φαίνεται να το δεχτεί το Συμβούλιο θα θέλαμε όμως να επιμείνουμε μια και είναι η κόκκινη γραμμή για την Επιτροπή Περιφερειών αυτό ακριβώς, μια ευληγησία ε, που, την οποία δεν θα πρέπει να παρνηθούμε. Και κάτι ακόμα σχετικά με το θετικό έλλειμμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού λόγω της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στις πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τις συνθήκες ε, δεν μπορεί να είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός μας αλλά τι θα γίνει αν αυτό σωρευτεί κάθε χρόνο που περνάει. Γι' αυτό συμμερίζομαι την απόψη του πρόεδρου Σούλτς που λέει ότι η τάση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί να εμφανίζεται και το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει κάτι και να την αποφύγουμε να διαγράψουμε οριστικά. Το Κοινοβούλιο επίσης διαφωνεί και έχει τη δική μας υποστήριξη για τη θέση του αυτή. Θα ήθελα να μιλήσω για ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα για την νομοθετική δέσμη τη πολιτική συνοχή και να δώσω συγχαρτήρια στη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Χούμπνερ ιδιαίτερα, για την επιτυχία της στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πολλέ από τις συμφωνίες με τα κράτη-μέλη ακριβώ, βλέπουμε ότι εμφανίζονται και στα δικά μας αιτήματα όπως η διατήρηση του κώδικα συμπεριφοράς ώστε να υπάρξει μια κατάλληλη διαχείριση στον όλο προγραμματισμό, στην όλη επεξεργασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων και επίση αναφορά των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ε, στο συνολικό πακέτο και τις προκλήσεις που υπάρχουν και σε περιφερειακό επίπεδο και οι προκλήσεις δημογραφικές ε, που να στα επιχειρησιακά προγράμματα. Και επίσης μια παρατήρηση. Μέσω αυτών των παρατηρήσεων συμφωνήσαμε το κοινό, με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό το μακροοικονομικό το ίσως να το δεχθούμε. Αυτό το 2014-2020 αυτό πολίτες πρόγραμμα έχει ορισμένες προϋποθέσεις ε, και θα πρέπει να δούμε την εκθέση του προπολογισμού και ταυτόχρονα την υποχρέωση των κρατών μελών από τη στιγμή που θα πρέπει να σεβαστούν τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαχείρισή τους στην οικονομική και τη φορολογική. Κάτι ακόμα να τονίσω κάτι το παράξενο εδώ για τις κυρώσεις, για τις ε, περιβολικά ελλείμματα. Ενώ προπολογούμε από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι έχει ακριβώς ένα διαφορετικό έλλειμμα. Ε, αυτό βλέπουμε και το οποίο θα αυξάνεται κάθε χρόνο που θα περνάει. Ζητάμε περισσότερη συνοχή λογική πάνω σε αυτό και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίζει να υποστηρίζει τις θέσεις του στον τριμερή διάλογο από τη στιγμή που θα ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Και εμείς είμαστε κατά το αποθεματικό απόδοση εθνικού 7% στο σύνολο των χρημάτων και για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αυτοδίακή. Και θα πρέπει να δούμε τις αρχές επί της διαχείρισης να, έχουν, να θέσουν στόχους εύκολους για να έχουν επιπλέον χρήματα. Εμείς προτείνουμε ένα απόθεμα ευέλικτο με να δούμε το πώς θα υποστηρίξουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Να πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ασχολήθηκαν ακριβώς με το πώς θα δίνουν τα χρήματα στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως και τις οροφές που θα ισχύουν. Και θα πρέπει να δούμε ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τι θα γίνει με μια υποχρεωτική διαβούλευση βέβαια της δικής μας Επιτροπής Περιφερειών. Αλλά δεν υπήρξε καμία σχετική νομοθετική πρόταση θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο γενικό κανονισμό. Και ακόμα κάτι σύντομα να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της περιφερειακής γενικά ανάπτυξης. Ο Γιώργος Όλμπριχτ πρότεινε να υποστηρίξουμε αυτή τη βάση με μια στενή συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω τον κύριο Όλμπριχτ για την πρότασή του και θα ήθελα να την υποστηρίξετε γιατί διαφορετικά θα ήταν αρνητικό να έχουμε νέες πολιτικές βάσεις ε, στα πλαίσια του 2020 και θα θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό. Και επίση παρακαλώ προσέξτε κάτι ακόμα για τη δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο διεθνού συνεργασία με τρίτες, σε τρίτες χώρες καλό θα ήταν να επιφέρουμε αλλαγέ στο νομοθετικό κείμενο. Αυτή τη μέση τη οικονομική κρίση, οι προκλήσει για την πολιτική συνοχή, για τις πολιτική συνοχή δεν ε, ήταν ε, πάρα πολύ μεγάλε. Και τώρα που θα πρέπει να ενισχύσουμε τι σχέσει μα με άλλου στον κόσμο για να πετύχουμε λύσει για κοινά προβλήματα που μα ταλανίζουν. Και εδώ από την Επιτροπή περιφερειών θα θέλαμε να ζητήσουμε από την εισηγήτρια να συμπεριλάβει τις σχετικές αυτές απόψεις στα όσα θα προχωρήσουν στον τριμερή διάλογο. Αυτά είναι κυρίε και κύριοι μερικά από τα σημαντικά για μας σημεία. Ο κατάλογος θεμάτων σημαντικών που θα πρέπει να ασχοληθεί κανείς στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων είναι ιδιαίτερα ευρύ, αλλά να περιστούμε στα σημαντικά θέματα και να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες συμφωνήσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο οικονομικής κρίσης ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα πρέπει να βλέπει και μακροπρόθεσμα τα πράγματα για να πετύχουμε τα κατάλληλε λύσεις ε, στα πλαίσια τη στρατηγική του 2020 και μια σωστή διαχείριση, διαχείριση στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά πολύ καλά σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Με την αρχή αυτή δεν θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς ε, ταυτόχρονη μεταφορά και χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Εμείς ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να υπερασπιστεί τις θέσεις του σύμφωνα με τις συνθήκες και να υπερασπιστεί τη θέση του απέναντι Συμβούλιο για τους πολίτες, για τις περιφέρειες της Ευρώπης, για τους Δήμους της Ευρώπης. Είναι δικοί μας πολίτες. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Η πρόεδρος. Συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβω τώρα. Έχουμε 6 με 7 εγγεγραμμένου ομιλητές στον κατάλογο. Να δηλώσετε τώρα αν θέλετε για να μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο χρόνο μπορούμε να δώσουμε στον κάθε ομιλητή. Ο Δαρή, ο πρώτος ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βαλκάρθαλ για την παρουσίασή σας. Να υπενθυμίσω αυτά που είπε ο χθε στην διάσκεψη των Προέδρων. Το ανώτατο όριο δαπανών που προέκυψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον προπολογισμό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν βελτιωθούν κάποια ποιοτικά στοιχεία του προπολογισμού. Διότι από ποσοτική πλευρά το Συμβούλιο βέβαια έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα ανώτατα όρια ε, εφόσον δεν έχουμε δικούς μας ε, ίδιους πόρους και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επηρεάσει. Αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε την ποιοτική πλευρά. Υπάρχουν ε, πολλά σημεία που συμφωνούμε με την Επιτροπή Περιφερειών όπως είναι η τροποποίηση των προοπτικών, η, η ευληγησία και ξέρουμε ότι για ορισμένα θέματα χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο και θέλουμε επίσης να μπορούν να μεταφέρονται από τις διάφορες κατηγορίες ε, οι πιστώσεις και να υπάρχει και η ε, αυτόματη μεταφορά των πληρωμών από τη μία χρονιά στην επόμενη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα κύριε Βαλκάρθελ και για το οποίο εργαστήκαμε από κοινού όταν εκπονήσαμε τις προτάσεις μας για τις ε, δημοσιονομικές ε, προοπτικές είναι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και στην, ε, στο ψήφισμα Σούρε και στο ψήφισμα Κάλφιν Μπέγκε που ενεκρίθησαν με πάνω από 70% των ε, βουλευτών και στη δική σας πρόταση για το νομοθετικό πακέτο για τη συνοχή αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει εκπεφρασμένη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της περιφερειακής πολιτικής και τα μακρονομικά, μακροοικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα ενός κράτους μέλους. Και με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η σύνδεση, θα τιμωρήσουμε τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιφερειών να διατηρήσουμε τη γραμμή μας. Και ελπίζω ε, στις απαντήσεις σας να μας πείτε πιο συγκεκριμένα εάν εμένει στη διατήρηση αυτής της σύνδεσης η Επιτροπή Περιφερειών. Φάνη Στελρόιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έχετε μια πολύ καλή συνεργασία τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Ε, υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί, οι δημοσιονομικές προοπτικές και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Όπως είπε ο κ. Γκαρίγα, η ομάδα μας ε, δεν μπορεί να ε, συνεχίσει με αυτές τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών. Έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο ε, και πρέπει οπωσδήποτε να μέσα στα πλαίσια του τριλόγου να υπάρξει μια διόρθωση αυτής της τάσης. Υπάρχουν οι διάφορες φάσεις ε, της διαδικασίας που δεν θέλω να επαναλάβω. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτό το πλαίσιο είναι 7 ετές. Αυτό είναι σαφές ε, υπήρξε σαφές μέχρι τώρα και πρέπει να, τηρηθεί αυτός ο στόχος ό,τι συζήτηση και να γίνει στο Κοινοβούλιο δεν πρέπει να τεθεί να αμφιβόλω αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική ε, και για μένα αυτό αποτελεί τη βάση ε, πολλών συζητήσεων. Ε, οπωσδήποτε υπάρχει ε, κάποια κριτική ε, που πρέπει να γίνει αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να, ζητήσω, να ρωτήσω την Επιτροπή Περιφερειών να δει αυτό το 7 ετές πλαίσιο. Ελπίζω ότι μέσα σε τρεις μήνες θα περατωθεί η παρούσα διαδικασία και όλοι οι συγητές θα μπορούσαν μαζί με τον Πρόεδρο να συζητήσουν το θέμα και με την Ιδανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δουλέψουμε σωστά, ούτω ώστε να έχουμε νέα μέτρα συνοχής για τις περιφέρειες. Και υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Βλέπω ότι εσείς ε, έχετε μηχανισμούς ελέγχου ε, παραδείγματος χάρη και ότι δράσατε, ε, δουλέψατε σωστά. Τώρα παραδείγματος χάρη έχετε να αντιμετωπίσετε μια μεγαλύτερη εξειδίκευση και πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμός όλων των οργάνων που έχουμε για την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχουν νέες προοπτικές για νέες δράσεις που πρέπει να τις ακολουθήσουμε, πρέπει να συγκεντρωθούμε, ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, τεχνολογία της ε, επικοινωνίας και ε, στην παρούσα περίοδο υπάρχουν μια καινούρια δυνατότητα εφαρμογών. Πρέπει να δούμε πώς θα υιοθετηθεί αυτή η καινούρια πολιτική στην, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των περιφερειών με μια επιπρόσθετη διάσταση γιατί υπάρχουν ορισμένοι που δεν ανήκουν βέβαια σε αυτή την Επιτροπή αλλά ανήκουν γενικότερα στο Κοινοβούλιο πιστε, ε, αναρωτιούνται σε τι χρησιμεύει η ύπαρξη της Επιτροπής Περιφερειών βεβαίως έχει ε, την ευθύνη την τελική το Κοινοβούλιο αλλά ο ρόλος ε, στην, για την εκπόνηση της περιφερειακής πολιτικής. Ο, ο ρόλος μας είναι να προσεγγίσουν τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους και βέβαια να έχουν και κάποια σχέση με το εκλογικό σώμα εν ώψη των εκλογών του επόμενου έτους. Νομίζω ότι χρειάζεται, χρειάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και ένας έλεγχος, όχι νέος έλεγχος, αλλά καλύτερος έλεγχος. Ίσως ε, μέσα στους επόμενους μήνες θα πρέπει να παρέμβω από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, μας είπατε πως έχει κατάσταση και σίγουρα συμφωνούμε μαζί σας ε, ότι ε, αυτή η συμφωνία σε αυτό το πολιετές πλαίσιο του Συμβουλίου δεν ε, είναι εκείνη που θα απαιτούσε κανείς τα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ε, για το 2020. Εσείς η Επιτροπή Περιφερειών ε, θα πρέπει να χτυπήσετε το κουδούν του κινδύνου ακριβώς ε, πάνω σε αυτές τις προκλήσεις. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε τρία σημεία. Η πρώτη πρόκλησή μας είναι της κλιματικής αλλαγής και ενεργειακή πολιτική. Να υπενθυμίσω κάτι ότι όλη η συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος από τη βάση θα ξεκινήσει όχι από τις πόλεις, ε, όχι από τις περιφέρειες. Όλες αυτές οι πηγές οι ενεργειακές αποτελούν πρόκληση γιατί δημιουργούν και άλλα θέματα και προβλήματα όπως την επαναβιομηχανοποίηση της οικονομίας ε, επιτόπου και να έχουμε μια πραγματική διαχείριση και εσείς θα πρέπει να μιλήσετε για αυτή την μεταβατική περίοδο για να μπορέσουν και οι επιτόπου φορείς να παίξουν το ρόλο τους. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Και η δεύτερη τώρα, το είπατε, είναι η οικονομική πρόκληση με τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τις ανεργίες, την ανεργία Υπάρχουν χώρες που έχουμε και 60% ανεργία νέων και εκεί θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να παίξει εκεί επιτόπου ρόλο η οικονομία και μάλιστα έξυπνα πάνω σε νέους τομείς και πράσινους τομείς. Η επόμενη πρόκληση είναι η κοινωνική οικονομικές προκλήσεις ακριβώς ε, να αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια τόπου Βλέπουμε τώρα και περισσότερο ε, ασκείται μια διάκριση να με την περιοχή και την πόλη και υπάρχουν ε, αδικίες απαράδεκτες και λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να παραμείνει απαθές θα πρέπει να υπερασπίζει πάντα την αρχική του θέση να απορρίψει αυτή τη συμφωνία και να δείξει ακριβώς και το Κοινοβούλιο και το Επιτροπή να συνδυαστούν, να συνεργαστούν καλύτερα για να προετοιμάσουν μια συμβαστική λύση. Με ανησυχεί η σημερινή κατάσταση. Για ποιο λόγο βλέπουμε ότι προχωρούν αργά-αργά τα πράγματα στη πραγματεύση και στον τριμερή διάλογο εμείς βλέπουμε τι γίνεται με την μελλοντική πολιτική συνοχής ε, και το Συμβούλιο πάντα αναποφάσιστο είναι καθυστερεί στα σημεία κλειδιά της συμφωνίε. Και εσείς χρειάζεστε όμως απαντήσεις ε, και για τις περιφέρειες που θέλουν να δουν το θέμα της συγκέντρωσης εκεί και νέες περιοχές που θα ενταχθούν σε μια κατηγορία, είναι αυτές οι σε μετάβαση κατηγορίες ε, και να δούμε τα κύρια σημεία σχετικά με αυτά τα θέματα για να προχωρήσουμε από νωρίς νωρίς ε, και ακόμα σε αυτή την κρίσιμη καμπή δεν τα αντιμετωπίσαμε. Είναι όμως καθοριστικά για το μέλλον σημεία Να σας πω ότι σίγουρα αν δεν προχωρήσουμε με ένα φιλόδοξο προπολογισμό και μια κατάλληλη αντιμετώπιση που είναι αντίστοιχη με τις προσδοκίες, τότε θα είναι καταστροφικό για τις περιφέρειες αυτές. Για ποιο λόγο. Απλά και μόνο αυτό που κάνουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι κάνουμε. Προσπαθούμε να προλάβουμε. Αλλά και εσείς θα πρέπει να προλάβετε τι όμως τις προσεχείς εταιρικέ συμφωνίες, τα επιχειρησιακά προγράμματα και όσο καθυστερεί κανείς, τόσο καθυστέρηση θα υπάρξει στον επόμενο προγραμματισμό, στο ξεκίνημά του. Εκεί είναι το δραματικό της καταστάσεως, γιατί δεν θα είμαστε έγκαιρα έτοιμοι. Άρα λοιπόν, το μήνυμα της Επιτροπής Περιφερειών σήμερα γιατί αυτό το μήνυμά σα εδώ στην Επιτροπή μας, ε, στην Επιτροπή μας Περιφερειακή Ανάπτυξη δεν θα πρέπει να ακουστεί μόνο από τη δική μα Επιτροπή, αλλά από το Κοινοβούλιο στο σύνολό του και κυρίως από το Συμβούλιο. Εσείς τώρα πώς θα ενεργήσετε ώστε το μήνυμα σας αυτό να ακουστεί. Πάντως είναι το ίδιο μήνυμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο ένας δίπλα στον άλλο να προχωρήσουμε για ένα φιλόδοξο προπολογισμό με καλό συλλογισμό και κυρίως για τους ίδιους πόρους για τον προπολογισμό και θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η Ευρώπη γιατί η Ευρώπη ε, ακριβώς δεν θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα λιτότητας επιτόπου. Έχουμε ακόμα 7 άτομα που θα πρέπει να λάβουν το λόγο. Γι' αυτό σας παρακαλώ όσο γίνεται συντομότερα. Πάμε Α, ναι, για να συμπληρώσω. Μας είπατε μισόδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Α, δεν είναι κατάλληλη έκφραση. Στο Συμβούλιο, βλέπω από όσα έγιναν ε, πριν από λίγο, μια ρήξη ιστορική μπορώ να πω. Πρώτη φορά είναι που οι ευρωσκεπτικιστές επικράτησαν στον όλο μηχανισμό οικοδόμησης της Ευρώπης. Ρήξη λοιπόν που μας ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί όλοι υποστηρίζουν πια τον Κάμερον και την ε, Βρετανική κυβέρνηση με τον τρόπο, βρίσκουν τις κατάλληλες ε, δικαιολογίες και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει ιδιαίτερα να αντιδράσουν ε, ακόμα και σε πλαίσια μιας κρίσης στους χώρους αυτούς γιατί χωρίς μια παρόμοια αντίδραση γιατί ακριβώ ε, έτσι εξηγείται όμω και αυτή η επιστοδρόμηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών κυβερνήσεων. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα και με τα όσα έχει διάθεσή του από την ε, συνήθεια δεν θα πρέπει να συμμετάχει, αλλά θα πρέπει να... Νίκο, έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα στο Κοινοβούλιο θέλουμε να προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι ένα από τα εργαλεία εφαρμογής και επίτευξης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είτε αυτό αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, είτε τη συνοχή, είτε την απασχόληση των νέων, είτε τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής ή της κοινή ελευτικής πολιτικής. Άρα πρέπει να εξετάσουμε τον προπολογισμό από δύο οπτικές. Κατά πόσο είναι, ε, είναι επαρκής η της κοινη ελευτικη πολιτικης αρα πρεπει να εξετασουμε τον προπολογισμο απο δυο οπτικες κατα ποσο ειναι ειναι επαρκης η πορη που διαθέτει, αλλά και κατά πόσο βοηθάει στο να υλοποιήσουμε τέτοιες στρατηγικές. Πολλές φορές δαπανούμε τεράστια ποσά και χωρίς όμως αυτό να έχει ένα αποτέλεσμα πάνω στην βελτίωση της ζωής των πολιτών, την αναζωγόνηση της οικονομίας ή την απασχόληση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο ποστό ανεργίας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πόροι που θα διατεθούν για τους νέους με το κριτήριο των περιοχών που έχουν πάνω από 25% ανεργία θα είναι 6 δισεκατομμύρια αν το μοιράσουμε αυτό με τον αριθμό των ανέργων νέων σήμερα στην Ευρώπη, που είναι πάνω από 8 εκατομμύρια, αντιστοιχούν 750 ευρώ για να κάνουμε πολιτικές για την απασχόληση των νέων ανά νέο σε διάστημα 7 χρόνων. Να συγκρίνουμε αυτό το ποσό με 100 δισεκατομμύρια για να διασώσουμε το τραπεζικό σύστημα. Αλλά πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες το 2014 ότι πρέπει να ψηφίσουν σε ευρωεκλογέ όταν το ποσό που αντιστοιχεί για την πολιτική για του νέου είναι απειροελάχιστο. Εάν επενδύαμε πραγματικά όπω πρέπει να είναι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα και στο θέμα τη οικονομία και στα θέματα τη κοινωνική συνοχή θα ήταν πολύ καλύτερα. Σα φέρω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα για να διασωθεί θα χρειαστεί 240 δισεκατομμύρια. Είναι το 1 τέταρτο του προπολογισμού που συζητάμε σήμερα για 7 χρόνια για όλη την Ευρώπη. Όμως από αυτά τα χρήματα τίποτα δεν πάει πραγματικά στην αναζωογόνηση οικονομίας και στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Απλώς, εάν διατηρούσαμε σε ένα επίπεδο την οικονομία, θα μπορούσαμε να έχουμε μειώσει το χρέος κατά 20%, όπως λένε οι οικονομολόγοι. Άρα είναι σωστό όταν λέμε να διαθέτουμε τα χρήματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με πιο σωστό τρόπο, αλλά αυτό πρέπει να το συζητάμε πράγματι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ορισμένοι το εννοούν για να περικόψουν τον προπολογισμό, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, την κρίση που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για του Απόρου, το οποίο έχουμε στήσει και εδώ πέρα. Οι πόροι θα διατεθούν είναι 2,5 δι. Όταν έχουν πολλαπλασιαστεί οι φτωχοί, ο αριθμό των φτωχών σε όλη την Ευρώπη. Με 2,5 δι μπορούμε να κάνουμε πολιτικέ για του φτωχού. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Και τέλος να μην συγκρίνουμε τον προπολογισμό το κάνουμε πολύ συχνά και στο Κοινοβούλιο αλλά κυρίω εκτό Κοινοβουλίου, το πολιετε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 το συγκρίνουμε με την προηγούμενη περίοδο, 2007-2013. Όμω Όμως συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές. Αλλιώ φανταζόμασταν θα εξελιχθεί η οικονομία, η κοινωνική συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα αυτό ο προπολογισμό του 2014-2020 είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει αυτόν τον προπολογισμό, ο οποίο αφενό είναι ελληματικό, αφετέρου δεν κατευθύνεται στοχευμένα στο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, δηλαδή συντηρεί παλιά, παλιές προτεραιότητες, ενώ πρέπει να στραφεί σε καινούριε προτεραιότητες και πραγματικά δεν βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως είναι η ανεργία, όπως είναι η, η, η μεγένθηση της, ε, των διαφορών μεταξύ των περιφερειών, όπως και το γεγονός ότι σήμερα έχουμε περισσότερες φτωχές περιφέρειες στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πρέπει πραγματικά να αρχίσει σοβαρή διαπραγμάτευση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και να πάμε σε ένα προπολογισμό ο οποίο θα είναι πραγματικά ε, βοηθητικό τη πολιτική συνοχή τη περιφερειακή ανάπτυξη και θα είναι επενδυτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you, dear colleagues. We have... Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ήδη εξαντλήσει το χρόνο που έχουμε για αυτήν την απόψεων και υπάρχουν ακόμη πέντε ομιλητέ. Θέλετε να απαντήσετε τώρα, λέει η κυρία Χούμπνερ. Στον κύριο Βαλκάρθελ. Όχι, στο τέλος. Ωραία. Θα συνεχίσουμε τώρα τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι, να μην ξεπερνάτε τα ένα-δύο λεπτά, γιατί αλλιώς θα έχουμε δυσχέρεια. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Βαλκάρθελ, με αυτές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εντάξει, συμφωνούμε πάνω σε κάτι ότι δεν διαθέτει τα μέσα σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει τη μάχη της κατά της κρίσης και να έχουμε και πάλι ανακαμψή. Η περίοδη αυτή είναι μοναδική στην ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμών ιστορική στιγμή στην όλη ιστορία της περιφερικής πολιτικής. Γιατί πρώτη φορά στην ιστορία της περιφερικής πολιτικής που προτείνεται ένας μειωμένος προϋπολογισμός. Περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερος και σίγουρα μια μείωση δεν μας ικανοποιεί γιατί θα επηρεαστεί το σύνολο της περιφερειακής πολιτικής παρακαλώ προσέξτε κάτι. Στο 77 της απόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι αναφέρεται οι δυνατότητες οι μακροοικονομικές ε, όχι. Και στον τριμερή διάλογο προσπαθούμε να διατηρήσουμε όμως τη θέση αυτή απέναντι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και από τη στιγμή που διαπραγματεύομαι εγώ λέω γιατί αυτό το μακροοικονομικά οι δυνατότητες τι ρόλο για το περιθώριο ελιγμό το οποίο μας επιτρέπουν πια. Και παρακαλώ συνάδελφοι προσέξτε αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο μέσω της συναπόφασης ε, γράφουμε τα άρθρα των ε, εσωτερικών σχέσεων για τις δυνατότητες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντικότατο λοιπόν είναι διάφορες αρχές να μείνουν, παραμείνουν σεβαστές και να μην δεχτούμε να μας θέσουν μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. Δεύτερη παρατήρησή μου. Βλέπουμε σιγά σιγά πώς προχωράει η κατάσταση στους κανονισμούς ότι μπαίνουν εκεί ανάμεσα διάφορα στοιχεία τα οποία αλλάζουν τις ίδιες αρχές της περιφερικής πολιτικής και πριν έρθετε εσείς είχαμε μια συζήτηση για τις κρατικές ενισχύσεις που πάνε στις περιφέρειες και εκεί στις νέες ρυθμίσεις όπως τις βλέπουμε Υπάρχουν ε, έτσι παράξενα βλέπουμε ότι γλιστρούν εκεί ανάμεσα διάφορες ρυθμίσεις, ε, κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι για χώρες ε, της συνοχής. Και σε αυτό πάνω λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερα να υπαγρυπνούμε και να έχουμε όλοι μας συνειδητοποίηση ότι οι προτινόμενες συμβαστικές λύσεις δεν μας ικανοποιούν. Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε μια περιφερειακή πολιτική που είναι στο ύψος των προσδοκιών. Κάτι ακόμα. Είναι σημαντικά τα όσα θα γίνουν γιατί θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται να προσέξουμε να μην πούμε ακριβώς, να μην υποστηρίξουμε ότι ε, πάση θυσία πέραν τη διάφορες παραχωρήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε σαν κατάληξη μια συμφωνία. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει στη θέση του και να υποστηρίξει ότι είναι απαράδεκτος ένας παρόμοιος προϋπολογισμός. Κορνέλια Ευχαριστώ. Πολλά ήδη υπόθηκαν, αλλά να τα πω ακόμη πιο έντονα. Έτσι όπως διατυπώθηκαν οι δημοσιονομικές προοπτικές από τα πορίσματα του Συμβουλίου είναι αν να μην υπάρχει καμία προηγούμενη απόφαση για τα θέματα αυτά. Το Συμβούλιο αγνόησε πλήρως το Κοινοβούλιο. Όλα που είναι σημαντικά για μας ή τουλάχιστον τα περισσότερα που είναι σημαντικά για μας χαρμόσυνα τα αγνόησε. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει και από την Επιτροπή Περιφερειών ένα κατηγορηματικό 38 όχι. Να υποθεί σαφώς και από εσά όπως και από εμά ότι είναι απαράδεκτος. Γιατί θα ήταν παράνομος ένας τέτοιος προπολογισμό. Θα ήταν παράνομος διότι δεν είναι δυνατόν να είναι ελληματικός ο ενωσιακός προπολογισμό. Δεύτερον, ανεργία των νέων. Έξι δις. Γελίο ποσό. Γελίο το τονίζω. Θα έπρεπε στα διευθυντικά ταμεία να υπάρχει μια ειδική ρήτρα για τους νέους. Ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθούνται κατά προτεραιότητα μέσω των διαθροτικών πόρων. Και επιπλέον αυτά τα έξι δις τα βάζουμε από διάφορες, είναι συνοθήλευμα χρηματοδοτήσεων από διάφορα ταμεία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοια λύση. Και τελευταίο, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Βεβαίως την καταπολεμήσαμε, γιατί δεν έχει καμία έννοια. Είναι απλά και μόνο ένας τρόπος για να εμποδιστούν οι χρηματοδοτήσεις των περιφερειών. Θα πρέπει να είναι κόκκινη γραμμή μας αυτό. Και τελευταίο, τι θα πρέπει να κάνει τώρα το Κοινοβούλιο. Εάν θέλει επιτέλους να παλέψει, πρέπει να συμφωνήσει επί προτεραιοτήτων. Πού θέλουμε όλες τις πολιτικές ομάδες να τονίσουμε ότι δεν, διαφωνούμε, ότι δεν συμφωνούμε και πού μπορούμε να κάνουμε συμβασμούς. Και θα πρέπει να εμείνουμε περαιτέρω στο Συμβούλιο, όπως και τόσα πολλά χρόνια στο παρελθόν, να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Η Μαρία Ιρηγογέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε. Ε, εδώ άκουσα διάφορες απόψεις από διάφορα ε, Πολιτική ομάδε, αλλά δυστυχώ ε, δεν είμαι πλήρω ικανοποιημένο. Αυτό είναι απαράδεκτο αυτό ο προπολογισμό. Η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αυξάνει τον προπολογισμό τη. Ε, αυτό είναι ένα ποσοστό γελίο για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ε, εδώ δεν υπάρχει πια φιλοδοξία στο Συμβούλιο και δεν έχουμε πια εμπιστοσύνη στα πολιτικά μέτρα για την πολιτική οικονομία. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα μέτρα λιτότητας. Εσείς ε, εκπροσωπείτε τη Μούρθια που χάρη στην Ισπανία, που χάρη ακριβώς στις ενισχύσεις ας πούμε ξεπέρασαν τα προβλήματα του σεισμού εκεί. Αυτός ο προπολογισμό που να πούμε ότι είναι λογικός ε, είναι ένα προπολογισμό πολύ χαμηλότερος από το πολιτιών. το 12% του ΑΕΠ για τις ανάγκες αυτές να τις καλύψεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση για τους νέους. Εδώ για τον δείκτη του αναργίας αυτός δεν είναι μόνο για το ΑΕΠ αλλά για τη Μαδρίτα ας πούμε περιοχή που είναι πάνω από το 70% έχει παρόλα αυτά έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας παρακαλώ για σκεφτείτε το, ένας δείκτης, ένας δείκτης που δείχνει την πραγματικότητα. Εμείς εργαζόμαστε με προβλέψεις, θα πρέπει να δούμε όμως και τα σκηνικά, τα προβλέψιμα και θα πρέπει να δούμε ότι με την οικονομική αυτή πολιτική δεν θα πετύχουμε την επιθυμούμενη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Γιώση Ματούλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί δεν θέλω να επαναλάβω όσα ήδη υπόθηκαν. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συγκεντρωτικά και αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τις περιοχές, ιδιαίτερα στην ε, Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα στη χώρα μου, τη Ρουμανία. Πώς θεωρείτε ότι θα επιχειρήσουμε να υπάρξει περισσότερη εξισορρόπηση στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή να υπάρξουν εταιρικέ σχέσει με τα κράτη-μέλη και να διαχειριζόμεθα την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχή συγγνώμη, σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, ο ρόλο των περιφερειών πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και αν το πιστεύετε, πώ θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τι βήματα θα αναλάβετε προ αυτή την κατεύθυνση για να σα υποστηρίξουμε ευχαριστώ. Γιάννη Όλμπριχτ. Υπάρχουν διαφορετικές ε, ερμηνείες. Ε, άκουσα ότι εσείς προτείνετε να ε, μπλοκάρουμε τη συμφωνία αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είχα κατανοήσει έτσι τα πράγματα. Αν είχα, εγώ είχα καταλάβει ότι ε, θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτά που μοιραζόμαστε, ε, την ευελιξία μας και τις διάφορες αρχές που απαριθμίσαμε. Θέλω να διευκρινίσω λίγο την κατάσταση, γιατί ε, δεν θέλω να έχει έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή Περιφερειών για να υποστηρίξει πιο ακραίες θέσει του Κοινοβουλίου σε τελική ανάλυση. Ε, η μία, ένα από τα προβλήματα είναι το θέμα του ελλείμματο που το είδαμε εδώ με μεγάλη σαφήνεια. Πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικά στοιχεία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ένα είναι ε, η, το, το έλλειμμα το 12 και το 13, η τρύπα που η λεγόμενη στον προπολογισμό. και το άλλο είναι η ανάληψη υποχρέωση για πληρωμέ. Και εδώ είναι ε, μια δεκαετή προοπτική ενώ οι πληρωμές υπάρχουν για 7 χρόνια και θα χρειαστούμε επιπρόσθετα άλλα 3 χρόνια για να μπορέσουμε να πληρώσουμε το χάσμα που θα υπάρξει μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών και ε, θα πρέπει δηλαδή να αγωνιστούμε για μια καλύτερη κατάρτιση του προϋπολογισμού ίσως να πρέπει να αναθεωρήσουμε την δημοσιονομική πολιτική ε, μακροπρόθεσμα γιατί ήρθε η κατάλληλη στιγμή τώρα αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνουν ένα-ένα ε, και θέλω να υποβάλω και μια παρατήρηση. όταν αρχίσουμε τον τρίλογο έχουμε ένα ε, ε, στοιχείο για τις ε, τοπικές ε, αρχές και τις περιφερειακές αρχές άμεσα για τις λεγόμενες για τις μεγάλες πόλεις για τις μεγάλες αστικές περιοχές το Συμβούλιο είναι κατά οι περιφερειακές αρχές δεν θέλουν να δώσουν να κάνουν καμία υποχώρηση σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ε, αστικές περιοχές και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Επιτροπή Περιφερειών και ελπίζω να μας βοηθήσετε να το λύσουμε γιατί εμείς μαχόμαστε για την, για την εκχώρηση αυτή ενώ το Συμβούλιο είναι ανοιχτά εναντίον. Ε, ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής ο κύριος Ούγκια. Πρόεδρε ευχαριστώ. Με εκπλήσει πραγματικά η υποστήριξη του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών στον προϋπολογισμό. Πολλές φορές δώσαμε κοινή μάχη εδώ. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ειδική οπτική για τις περισσότερο μειονεκτικές περιοχές στα πλαίσια της Περιφερειακής Συνοχής. Και πολλές φορές είχαμε από την Επιτροπή Περιφερειών προτάσεις που βελτίωναν τα πράγματα. Γι' αυτό εκπλήσωμαι. Τώρα που άκουσα τα λόγια σας ε, επιβεβαιώνεται αυτό το αρνητικό που θα δοθεί από τους φιλελεύθερους ε, την αρνητική ψήφο, γιατί είναι αρνητικός ο προπολογισμός που δεν είναι υπέρ της ανάκαμψης οικονομικής, είναι ακόμα περισσότερο εις βάρος των περιφερειακών και μειονεκτικών περιοχών παίρνουν ένα νόημα εδώ σε θεσμικό επίπεδο αυτά τα λόγια. Να σας απευθύνω μια ερώτηση συγκεκριμένη, απλή, ακριβή. Το Επιτροπή Ελευθεριών, τι γίνεται τις νησιώτικες περιφέρειες ε, και το ξέμα των προβλημάτων, πώς θεωρεί θετικό ή αρνητικό τον προπολογισμό. Εσείς μιλήσατε θετικά για τον προπολογισμό αυτόν. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, έχετε τον λόγο. Ωραία. Καταρχάς ευχαριστώ όλους όσους πήραν τον λόγο διότι η συζήτηση που έγινε μου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω κάποια θέματα που ίσως δεν ήταν σαφή ευθύς εξ αρχής δεύτερον να τονίσω ότι η Επιτροπή Περιφερειών στην οποία συμμετέχω εδώ και 18 χρόνια αλλά ίσως επειδή έχω 18 χρόνια μέλος της ξέρω πολύ καλά ποια είναι η φύση της Επιτροπής Περιφερειών. Η Επιτροπή λοιπόν Περιφερειών έχει κάποια όρια στη δράση της, δεν έχει καμία νομοθετική αρμοδιότητα, καμία απολύτως, απλώς εκπονεί εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις που έρχονται σε εσά εδώ και τις οποίες εσείς εξετάζετε και μπορεί και να τις απορρίψετε. Αλλά παρόλα αυτά τις εκτιμάτε. Πιστεύω ότι οι περισσότερες εκθέσεις μας αξιοποιούνται και νομίζω ότι πολλές φορές μια έκθεση που ξεκινάει από την Επιτροπή Περιφερειών γίνεται νόμος μέσω του Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση. Η σχέση είναι ευέλικτη, αλλά γίνεται όλο και πιο στενή αυτή η σχέση ανάμεσα σε εμά και σε εσά. Αλλά έχω κάθε συνέστηση ότι έχουμε το ρόλο μας εμείς ως Επιτροπές Περιφερειών και κατέχουμε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά τίποτα παραπάνω. Να είναι λοιπόν σαφές αυτό. Δεν νομίζω ότι είπα, καθόλου μάλιστα, κατά την ομιλία μου, ότι θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο είναι θετικός. Νομίζω ότι υπήρξα σαφής. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ πολλές φορές, ούτε να το εξηγήσω. Γιατί δεν το είπα. Δεν είπα καμιά στιγμή στην προηγούμενη ομιλία μου δεν χρησιμοποίησα τον όρο θετικός ο προπολογισμός. Γιατί αντίθετα δεν είναι θετικός. Είπα ότι περιέχει μεγάλες περικοπές, μεγάλες ελλείψεις. Και τονίζω μεταξύ αυτών ότι μπορεί κανείς να είναι σχετικά λογικά ικανοποιημένος εάν καταλάβουμε ότι υπάρχουν τρεις σαφείς συμπτώσεις μεταξύ της ε, θέσης του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών μακροοικονομική ρεσιμότητα απόλυτα συμφωνούμε ευληγησία απόλυτα συμφωνούμε και αποθεματικό εθνικής αποδοτικότητας για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το τρίτο αυτό θέμα. Και εδώ επίσης συμφωνούμε απόλυτα με το Κοινοβούλιο. Οπότε είμαι σχετικά λογικά ικανοποιημένος, διότι σε τελευταία ανάλυση συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπου, όπως επαναλαμβάνω, ευτυχώς η Επιτροπή Περιφερειών συμπίπτει με τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αν θέλετε να πω και περισσότερα. Διότι όπως ξέρετε είμαι από τους πολιτικούς που του αρέσει να τα λέει στα ράτα. Πέρα από την άποψη της Επιτροπής Περιφερειών είναι και η δική μου άποψη. Συμφωνώ απόλυτα με τις πλευρές αυτές που προτείνει η Επιτροπή Περιφερειών και οι οποίες συμπίπτουν με τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει λοιπόν η ικανοποίηση ούτε προσωπική ούτε συλλογική ούτε θετικά στοιχεία του προπολογισμού. Υπάρχει σχετική ικανοποίηση επειδή συμπίπτουμε και πολύ στενά μάλιστα απόλυτα επιθεμάτων που κατά τη γνώμη μου είναι ζωτικά εάν θέλουμε να επιτευχθεί ένας προπολογισμό ή τουλάχιστον κάποια κριτήρια για την εκπόνησή του. Θα ήταν επίσης ε, λογικό να τονίσω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει ο προπολογισμό μόνο λόγια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ σας λέω εγκρίνεται τον προπολογισμό όπως ακριβώς τον παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι, όχι. Καθόλου μάλιστα το αντίθετο. Νομίζω ότι είπα σαφώ. όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είπα, ότι ο προπολογισμό ως διαδικασία δεν έχει λήξει. Έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του και είπα ακόμη περισσότερα πράγματα. Τώρα αρχίζει η διαδικασία του προπολογισμού γιατί τώρα ήρθε η σειρά του Κοινοβουλίου. Προηγουμένως ήταν η σειρά της Επιτροπής να παίξει το ρόλο της. Μετά ήταν η σειρά του Συμβουλίου. Τώρα ήρθε η σειρά του Κοινοβουλίου. Έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησα την ομιλία μου. Τώρα το Κοινοβούλιο πρέπει να του δώσει την οριστική του μορφή. Και αυτό σας ζήτησα. Και παραλαμβάνω. Δεν πρέπει να θίξουμε τις προοπτικές μας. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη στις περιφέρειες και τους πολίτες, να τους αφήσουμε όλους αυτούς χωρίς ένα σημαντικό όργανο ανάπτυξης όπως είναι ο προπολογισμό και οι προοπτικές, οι οποίες έχουν ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο, 7 ετές και συνέχισα λέγοντα ότι δεν πρόκειται να εγκρίνουμε αυτόν τον προπολογισμό. Πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Να επιδιώξουμε, να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το Κοινοβούλιο να αποδείξει τη δύναμή του που την έχει. Ούτω ώστε ο προπολογισμό να μεταβληθεί, ούτω ώστε να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε των πολιτών. Κοιτάξτε, έξω κάνει πιο κρύο από εδώ μέσα. Και αυτό ισχύει και για του ευρωβουλευτές και για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τους προέδρους των περιφερειών και βεβαίως και για τους δημάρχους και οποιουσδήποτε άλλους τοπικά εκλεγμένους ή γενικά εκλεγμένους. Οι απλοί άνθρωποι την περνάνε πολύ δύσκολα. Και είναι σαφές ότι πρέπει εσείς να τους βοηθήσετε να διαπραγματευτείτε με την στεναρότητα που σας χαρακτηρίζει, ούτω ώστε να καταλήξετε στο τελικό στόχο, ο προπολογισμό να είναι μέσο ανάπτυξης για την Ευρώπη. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Και επίσης είναι και γραμμένο. Οπότε μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Μπορείτε να το δείτε. Και υπάρχουν και γραπτά κείμενα. Υπάρχει μια απόλυτη αντίφαση. Να λέγεται ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό ή μάλλον το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να λέγεται λοιπόν από τη μία ότι είναι το μεγάλο όργανο ανάπτυξης που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξέλθει από την κρίση και παράλληλα να μην θέλουμε να ξεπεράσει το προηγούμενο που εξακολουθεί να ισχύει. Αντίθετα να αποτελεί μείωση μέσω των περικοπών. Δεν έχει έννοια. Είναι ψέμα να λέγονται αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Είναι αντίφαση. Και το είπαμε, το τονίσαμε. Το είπα προσωπικά και το παραλαμβάνω. Και θα το πω πολλές φορές ακόμη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει τώρα είναι να βελτιωθεί ό,τι είναι βελτιώσιμο. Και αυτό σας ζητώ να κάνετε. Και δεν το λέω προσωπικά, γιατί δεν είμαι εδώ παρόν προσωπικά. Εκπροσωπώ την Επιτροπή Περιφερειών. Και η Επιτροπή Περιφερειών θέλει να βελτιωθεί αυτός ο προπολογισμό. Αλλά παράλληλα η Επιτροπή Περιφερειών οποτεδήποτε είχε την ευκαιρία να το κάνει, πάντα είπε ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μείνουμε χωρίς προϋπολογισμό. Διότι οι περιφέρειες μας, οι τοπικές αρχές χρειάζονται αυτούς τους πόρους για να προσπαθήσουν να υπερβούν την κρίση. Βεβαίως δεν είναι αυτός που χρειαζόμαστε. Πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Αλλιώ δεν θα τον εγκρίνουμε. Αλλά πρέπει να επιδιώξουμε, να επιτύχουμε τη δυσχερή ισορροπία ανάμεσα στο εφικτό από τη μία πλευρά και το επιθυμητό από την άλλη. Είναι θεμελιώδες αυτό. Δεν είναι αδύνατη αυτή η ισορροπία, αλλά είναι δυσχερέστατη. Αλλά οπωσδήποτε πιστεύω ότι οι απόψεις που σας παρουσιάζω ως Επιτροπή Περιφερειών είναι δεν μας αρέσει αυτός ο προπολογισμό. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες Ευρωβουλευτές, παρακαλώ βελτιώστε το. Και παράλληλα να επιχειρήσουμε με κάθε μέσο να μην μείνουμε χωρίς προπολογισμό. Διότι τότε θα έχουμε εμποδίσει κάθε προσπάθεια ουσιώδους προγραμματισμού υπέρβασης της κρίσης. Βεβαίως, η μακροοικονομική ρεσιμότητα είναι μια επιπλέον επιβάρηση για τις περιφέρειες, όπως το είπαν ορισμένοι ομιλητές. Γι' αυτό το λόγο απαιτούμε ελαστικότητα ως Επιτροπή Περιφερειών. Απορρίπτουμε πλήρως ένα αρνητικό εργαλείο που μπορεί να είναι και θανατηφόρο για, τα, για τις λογικές προσδοκίες των πολιτών. Αυτή η αρχή, η λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και διερωτώμεθα αν είναι καλό ή όχι να υπάρχουν νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Δεν χρειάζονται νέοι μηχανισμοί. Είπε ο κ. Φανίσταλροι ότι ε, περιπλέκεται η κατάσταση με τη δημιουργία άλλων νέων μέσων που θολώνουν την κατάσταση και μειώνεται η σαφήνεια της διαδικασίας επίτευξης των στόχων. Μα υπάρχουν ήδη, υπάρχει ήδη μία πλατφόρμα για την ε, παρακολούθηση, προώθηση των στόχων του 2020 και συνεργαζόμαστε αυτών των μηχανισμών με σας. Υπάρχουν ήδη μηχανισμοί και μπορούν να αξιοποιηθούν. Τώρα, η πιο σημαντική ερώτηση. Γιατί υπάρχει Επιτροπή Περιφερειών, εφόσον υπάρχει Κοινοβούλιο. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Αυτή είναι η αιώνια συζήτηση. Αιώνια. Ίσως πρέπει να τη συζητήσουμε ακόμη περισσότερο. Ορισμένοι λένε θα πρέπει τώρα εγώ να υπερασπιστώ την Επιτροπή Περιφερειών. Ε, βέβαια θα πείτε. Αφού είναι, Επιτροπή Περιφερειών, αφού είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, τι θα κάνει. Βεβαίω είμαι πρόεδρος. Αλλά είμαι πρόεδρος γιατί είμαι πρόεδρος μιας περιφέρειας της Ένωσης. Δεν θα μπορούσα να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών αν δεν ήμουν τοπικά εκλεγμένος. Υπερασπίζομαι δηλαδή ένα θεσμικό όργανο που το μόνο που κάνει είναι να ασκεί πολιτική ε, κοντά στους πολίτες. Πολιτική γειτονίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσεί δεν ασκείτε πολιτική γειτονία και εσεί το κάνετε. Εκλέγεστε από εκλογικέ περιφέρειες όπου πρέπει να κάνετε απολογισμό και των οποίων πρέπει να εκπροσωπείτε και να προωθείτε τα συμφέροντα. Αλλά θα ήταν παραλογισμός παράλογη ευγένεια να σα πω, κοιτάξτε, όλοι υπερασπιζόμαστε την ίδια γειτονία. Όχι, δεν υπερασπιζόμαστε όλοι τον ίδιο τρόπο, δεν είμαστε όλοι τόσο κοντά στου πολίτε. Κοιτάξτε, οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι τόσο κοντά. Ε, συγγνώμη, οι πρόεδροι των περιφερειών δεν είναι τόσο κοντά στους πολίτες όπως είναι οι, οι δημοτικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Επίπεδα ε, εγκύτητα στους πολίτες. Και το κάθε επίπεδο πολιτικής έχει το επίπεδο εγκύτητάς του. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχουν όλα αυτά τα επίπεδα. Διότι ορισμένοι θέτουν ερωτήματα όντας στην ουσία δίπλα στον πολίτη, πατώντας δίπλα του. Άρα υπάρχει διαφορετική εστίαση. Αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και περισσότερο συντονισμός. Να, αποφεύγονται επικαλύψεις. Εδώ υπάρχει θέμα συζήτηση. Και ευχαριστώ να την κάνουμε. Αλλά θα καταλάβετε ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ χρόνο. Δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε εσείς τον έχετε να μου το δώσετε, ούτε εγώ τον έχω. Γιατί ε, αν ε, μιλήσω λίγο περισσότερο θα χάσω το αεροπλάνο μου. Πρέπει λοιπόν να περιγράψουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Διότι ξέρετε ότι σήμερα θέτουμε μια σειρά από για να διευκρινίσουμε το πιο ευαίσθητο τμήμα της πολιτικής. Τι μας ζητάει ακριβώς ο πολίτης. Μιλάμε για μακροοικονομική ερεσιμότητα. Αλλά αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, ε. Αυτό που όμω το καταλαβαίνουν όλοι είναι πολιτικές απασχόλησης για παράδειγμα ή μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανέχειας ή κατά πολέμηση της κλιματικής αλλαγής γιατί υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά μεγάλη συνειδητοποίηση αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε όλα όσα κάναμε πριν διότι αν δεν υπήρχε το παρελθόν δεν θα ήμασταν τώρα στη θέση να συζητάμε αυτά που συζητάμε τώρα όλα είναι απαραίτητα αλλά σε αυτή την πολιτική εγκύτητας εμείς ως Επιτροπή Περιφερειών εργαζόμαστε για να εφαρμοστεί το λεγόμενο σύμφωνο των δημάρχων. Τι περιέχει αυτό και το λέω χωρίς καμία αλαζονία. Είναι το καλύτερο όργανο για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Για να υπάρξουν δεσμεύσεις υψίστης σημασίας για να υπάρξει ενεργειακή αποδοτικότητα. Ούτω ώστε λοιπόν να εφαρμόσουμε πολιτικές που όντω τις απαιτούν κατευθείαν οι πολίτες. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά αυτό το σύμφωνο των δημάρχων. Για μένα είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που έχουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που προκύπτουν από την κακή χρήση της ενεργείας, από την κλιματική αλλαγή το οποίο πολλοί αρνούνται ή πολλοί αρνούνταν ενώ τώρα κανείς δεν το αφισβητεί πλέον και η ενεργεία των νέων 6 δις γελίο ποσό το είπαν επανειλημμένα οι προηγούμενοι αλλά είναι 6 δις λέω ότι είναι καλύτερα από 0 δεν είναι μεγάλη μάχη και να πούμε ότι με 6 δις προσβάλλουμε τους νέους που δεν έχουν προοπτική αυτή τη στιγμή. Και αυτή η προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας των νέων είναι πολύ σημαντικό και οι εταιρικέ σχέσεις αυτό είναι. Μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε πολιτικές εγκύτητας, πολιτικές γειτονίες, πολιτικές που βοηθάνε ευρύτερα τις περιοχές. Και εδώ έχει η Επιτροπή Περιφερειών σημαντικό ρόλο να παίξει. Βεβαίως, θα κάνουμε την ετήσια συνέλευση των τοπικών οργανισμών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο βορρά και στο νότο της Μεσογείου και υπάρχουν σαφείς προσπάθειες εταιρική συνεργασίας όπως κάνουν προσπάθειες συνεργασίας και με τις ε, χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Και εδώ έχει σημαντικό ρόλο το... η Επιτροπή Περιφερειών. Ε, αναφέρθηκαν ορισμένοι στον ευρωσκεπτικισμό. Κύριε Αλφονσί, οπωσδήποτε είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό. Αλλά ξέρετε είναι και κάπως αναπόφευκτο. Εντελώς αναπόφευκτο. Όλα αυτά ξέρετε είναι κυκλικά φαινόμενα. Η Ισπανία όπως ξέρετε ε, έγινε μέλος της Ένωσης το 86. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτό σήμαινε ότι για πολύ χρόνο δεν συμμετείχαμε για κάτι που από κάθε άποψη γεωγραφική, ε, πολιτική, πολιτιστική ε, ήταν ε, φυσικό να είμαστε τμήμα του αλλά για λόγους της δικτατορίας δεν είχαμε καταφέρει να το κάνουμε πριν το 86. Με όλα αυτά θα έλεγα ότι δεν αισθάνομαι δεν αισθανόμουν καλύτερα ότι ήμουν πολίτης της Ευρώπης το 86 ενώ θα έπρεπε να είμαι. Αυτός ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι λοιπόν ε, κάτι το εντελώς καινούριο. Είναι κυκλικό φαινόμενο όπως και η κρίση. Όσο μεγαλύτερη είναι η κρίση, τόσο περισσότερος ευρωσκεπτικισμός θα υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι τον δικαιολογώ. Όχι καθόλου. Απλώς συμμερίζουμε την ανησυχία σας. Η ανησυχία όμως αυτή είναι κοινή σε όλους μας. Είναι μια ανησυχία που πρέπει να μας απασχολεί όλους, όλους τους υπευθύνου. Όλα τα πολιτικά όργανα. Από το δήμαρχο του πιο μικρού χωριού μέχρι τον πρόεδρο του πιο μεγάλου και ισχυρού κράτους της Ένωσης. Οπότε πρέπει να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων μας και παραλαμβάνω ο προϋπολογισμός όπως έχει τώρα δημιουργεί μεγάλες δυσχέρειες. Είναι πολύ δύσκολο να τον ε, υποστηρίξουμε, αλλά γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να κάνετε κάθε προσπάθεια και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας για να σας στηρίξουμε. Βεβαίως είναι τρομερές οι ε, περικοπές που γίνονται 30 δις, αλλά πρέπει και τα χρήματα να τα αξιοποιούμε καλύτερα και αποδέχομαι και την ευθύνη μου. Και πρέπει να απαιτήσουμε από όλους όσους διαχειρίζονται πόρους να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, καλύτερη δαπάνηση των πόρων. Είναι σαφές ότι έγιναν πολλά περίεργα πράγματα. Και τώρα είναι η ώρα να κλάψουμε. Είναι η ώρα να σκεφτούμε τα θέματα αυτά. Είναι θέμα τώρα να ψάξουμε να δούμε τι κάναμε λάθος στο παρελθόν. Κατά λίγο ε, ακούσαμε για την ε, ανεργία των νέων, την ε, μακροαιρεσιμότητα, τα είπαμε όλα αυτά. Ο ρόλος των περιφερειών θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ήταν η τελευταία ερώτηση. Ε, αυτή είναι η φιλοδοξία μας βεβαίως. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσε και σε μας μια μικρό, ένα μικρό άνοιγμα αν και ήταν μόνο η δυνατότητα ελέγχου της ε, επικουρικότητας. Αλλά προηγουμένως δεν το είχαμε. Είναι ένα μικρό έναυσμα. Είναι λοιπόν υπόθεση όλων μας. Και ημών, αλλά και ημών. Πρέπει η Επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειών ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν περισσότερη δυνατότητα αλλά και περισσότερη αποφασιστικότητα για να προωθήσουν ε, τις αρμοδιότητές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που με ακούσατε και για τις ερωτήσεις που μου κάνετε και ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση να μιλήσετε εδώ στην Επιτροπή μας και επίσης για τον πολύ ειλικρινή χαρακτήρα σας για το πώς συμμεριστήκατε όλα αυτά τα θέματα και της Επιτροπής Περιφερειών αλλά και ό,τι προέρχεται από την εμπειρία σας και την κατανόηση όλων αυτών των θεμάτων. Ε, εμείς μοιραζόμαστε τους στόχους μαζί σας. Είναι κοινή στόχη αλλά θα θέλαμε να σας δείξουμε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ε, τη δυνατότητα και τη βούληση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε στα χέρια μας έναν προϋπολογισμό και έναν καλό προϋπολογισμό για την Ευρώπη και για τις περιφέρειες της ε, με ανάπτυξη. Και ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, όλοι μας να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ ενός καλύτερου προϋπολογισμού και του να έχουμε έναν προϋπολογισμό στη διάθεσή μας. Είναι δύσκολο το εγχείρημα αυτό, αλλά αυτό προσπαθούμε να πράξουμε πράξουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Είμαι Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης αγαπητοί συνάδελφοι που είναι η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Καρόνα για την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον συντάκτη. Εδώ είστε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή για την κοινωνική στέγαση είναι κάτι το σημαντικό και ενδεικτικό γιατί αυτή η κοινωνική στέγαση βοηθάει και μάλιστα ιδιαίτερα για την επίτευξη διαφόρων στόχων της στρατηγικής ε, για το 2020 και για την ανάπτυξη και για το πόσο ελκυστικές είναι αυτές οι περιοχές αλλά και για τη μάχη κατά της φτώχειας και για την κοινωνική ένταξη. Όπως επίσης το πώς δίνει κανείς τη μάχη του απέναντι στα ενεργειακά προβλήματα και στις κλιματολογικές αλλαγές. Αυτά είναι σημαντικά. Από τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωτικό δεσμευτικό να εγγυώνται το δικαίωμα στη στέγαση. Επαναλαμβάνω λοιπόν για μας είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Για πολλούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να βρουν στέγη. Την περίοδο αυτή έγινε ένα στόχος ιδιαίτερα δύσκολος. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει ακόμα μόνιμη στέγη. Πάνω από το 18% επίσης ζούσε σε κατοικίες με πολλούς άλλους που δεν ήταν αξιοπρεπείς και πάνω από 10% επίσης ε, και αυτές οι εκτιμήσεις ε, είναι αρκετά χαμηλές δυσκολεύεται να αντέξει τα έξοδα του σπιτιού του. Άρα λοιπόν δυσκολίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο στέγασης. Και επειδή επιδεινώνεται η κρίση, επιδεινώνεται και το πρόβλημα. Γι' αυτό απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από δικής μας πλευράς να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι γίνεται, ό,τι μπορούμε μέσω και των διαρχοτικών ταμείων. Οι ανάγκες στέγασης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε ένα κράτος μέλος είναι διαφορετικές αυτές οι ανάγκες. Υπάρχει κάτι το σχετικό με την Δυτική Ευρώπη, κάτι διαφορετικό με την Ανατολική Ευρώπη και επίσης σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές και γι' αυτό όμως θα πρέπει να εγγυηθούμε ένα ενιαίο πλαίσιμο παρέμβασης. Γι' αυτό ακριβώς με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης έχουμε σαν στόχο να ευνοήσουμε μια παρόμοια πολιτική κοινωνική στέγασης ώστε όσο γίνεται περισσότερο να αξιοποιήσει για το 2014-2020 τα διοχετικά ταμεία σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την προστασία, την θερμική και τη χρησιμοποίηση ενός πηγών ενεργείας και επίσης την αηφόρο ανάπτυξη στην αστική και μία μάχη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Η γνωμοδότηση λοιπόν έχει κυρίως να κάνει με τα σημεία αυτά πώς τον προσεχή προγραμματισμό για επενδύσεις με προτεραιότητα για να μονώσουμε θερμικά καλύτερα τις κατοικίες και επίσης να βοηθήσουμε μια ανάπτυξη κυρίως σε μειονεκτικές περιοχές και να αποφύγουμε και απομονώσεις επικίνδυνες. Άρα λοιπόν δίνοντας μάχη υπέρ της κοινωνικής συνοχής και επίσης με επενδύσεις για την κοινωνική στέγαση στα πλαίσια σφαιρικότερων πολιτικών που να έχουν να επηρεάσουν θετικά τα πράγματα και σε πλαίσιο τοπικής οικονομίας με θέσεις απασχόλησης και κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και στήριξης μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν σημαντικός, ιδιαίτερα σημαντικός τομέας με προσπάθεια να δοθεί μία απάντηση από κοινωνικής πλευράς στα προβλήματα αυτά αλλά επίσης κάτι το επίσης σημαντικό να βοηθήσουμε την κοινωνική συνοχή και μια ανάκαμψη, μια αναθέρμανση της οικονομίας και με δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώχημ δεν είναι εδώ και ο δισηγητής, οπότε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδελφό μου ε, τον ε, κύριο Σαλβαδόρ Καρίνα για την εργασία του ε, ως συντάκτης της γνωμοδότησης ουσίας είμαι ικανοποιημένη από αυτή την εργασία συμμερίζομαι με τον συναδελφό μου τη βούληση που έχει να υπογραμμίσει τον ρόλο του μοχλού ε, της κοινωνικής στέγασης για να βγούμε από την κρίση και για, ως ένα νέο στοιχείο για την στρατηγική μας που είναι μια στρατηγική πρόοδου. Καταρχήν πρέπει να δούμε όλες τις θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία της απασχόλησης. Ε, το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το όφελος στην, σταθερότητα την μακροοικονομική. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προκαταλάβει αυτά τα θέματα με μακροοικονομικούς όρους ε, για την τεχνητή άνοδο των, ε, του στεγαστικού και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά όπως το, μας το υπενθύμησε ο συνάδελφος έχουμε την πάλι για την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να γίνουν τεράστιες επενδύσεις ε, ε, στο θέμα της μόνωσης, στο θέμα των ανανεώσιμων ενεργειών που πρέπει επειδή έχουμε καθυστέρηση να τις προωθήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Δηλαδή το πακέτο για το κλίμα ε, και κυρίως ο μεγάλος στόχος που είναι να μειώσουμε κατά το 1 τέταρτο τις εκπομπές των ρήπων μέχρι το 2000. 50. Ε, Επίσης, ο ρόλος ο θετικός της κοινωνικής κατοικίας είναι σημαντικός για την ε, συνοχή των περιφερειακών. Πρέπει να πω ότι για την διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα και για την προσέγγιση ε, στην πολιτική, στην κουλτούρα της συνοχής πρέπει να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οι οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς μοχλούς σημαντικούς έχει έναν πολιετή προϋπολογισμό μιλήσαμε για τη μάχη του προϋπολογισμού πριν από λίγο εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε τις επενδύσεις στα κοινωνικά ταμεία θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερα ποσά στη διάθεσή μας για να έχουμε καλύτερες επενδύσεις μαζικά η τελευταία ιδέα που θεωρώ πολύ σημαντική ως οικολόγος είναι ότι πρέπει πρέπει να υπερασπιστούμε ε, όλο τον τομέα που έχει σχέση με την ανάπτυξη των πόλεων. Υπάρχουν ορισμένες ε, ε, περιοχές μέσα στις πόλεις σήμερα που είναι προβληματικές και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της ανάπτυξης μέσα στο Ταμείο Συνοχής για την κοινωνική στέγαση για να βοηθήσουμε αυτές τις μειονεκτούσες γειτονιές. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να συνεργαστούμε με τον συντάκτη ε, της έκθεσης και επίσης ε, ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να υπάρχει από πλευράς Κοινοβουλίου μια επένδυση στην κοινωνική στέγαση που αποτελεί έναν από τους παράγοντες εξόδου από την κρίση που έχουν κατεπήγοντα χαρακτήρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Η στέγαση όντω είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι γίνεται μια συζήτηση σε αυτό το σημαντικό τομέα. Ωστόσο ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η στέγαση από την άλλη πλευρά είναι μια αρμοδιότητα εθνική, εθνική κυβερνητική ε, και είναι κάτι που πρέπει να επιληθεί ως πρόβλημα αυτό. Ε, πρέπει να, να υπάρχει μια αντίδραση σε, στο, σε πρώτο επίπεδο, στο πιο χαμηλό δυνατό επίπεδο. Συμφωνώ με την ε, προλαλή Πρέπει να... Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δράσουμε διαφορετικά. Χρειάζεται ένα ε, κέντρο... Ε, αλλά αυτό το κέντρο για το οποίο μιλάτε, κοινωνική στέγαση, θα δημιουργήσει μια περαιτέρω γραφειοκρατία. Ε, νομίζω ότι το, ε, υπάρχει η ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων και εκεί πρέπει να παραμείνουμε. Το θέμα της ενέργειας έχει διαφορετική σημασία για, του, για ε, τους ε, όσους προσπαθούν να επηρεάσουν παραδείγματο χάρη τις ενεργειακές τιμές για ορισμένους τομείς. Ε, είναι κάτι που πηγαίνει πολύ μακριά. Ε, εγώ έχω μια πολύ σύντομη παρατήρηση να υποβάλω. Ίσως θα πρέπει να εισάγουμε στο κείμενο μας ε, από πλευράς της Επιτροπής μας το θέμα των προβλημάτων που προκύπτουν όταν δεν έχουμε σαφή ορισμό του ε, εύρους της κοινωνικής στέγασης γιατί υπάρχουν εντελώς διαφορετικοί ορισμοί ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Έχουμε το περίφημο παράδειγμα της Ολλανδικής στέγασης που είχε ε, κρατικές επιδοτήσεις. Σε άλλα κράτη-μέλη επικρατούν διαφορετικές καταστάσεις. Ε, κοινωνική στέγαση για ορισμένα κράτη-μέλη σημαίνει ότι αφορά τους φτωχότερους, ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άλλους είναι, έχει σχέση με τους οργανωτές, τους ε, ιδιοκτήτες. Ε, το ΑΣΕΛΕΜ, δηλαδή ο Οργανισμός ε, ε, κατοικίας με φθηνή μίσθωση είναι τελείως διαφορετική στην Πολωνία από ότι είναι στη Γαλλία για παράδειγμα. Καλύτερα λοιπόν να καθορίσουμε το εύρος της στέγασης της κοινωνικής, το πεδίο ο κύριος Καρόνα θέλει να κάνει μια τελευταία, ένα τελευταίο σχόλιο ενδεχομένως. Ε, σύντομα, σύντομα. Με όσα ακούστηκαν συμφωνώ, ιδιαίτερα με το σχόλιο του συναδέλφου Όλμπρεχτ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ένας ορισμός ε, ομοιόμορφος μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν ε, ουσιαστικές βέβαια διαφορές, αλλά άλλο είναι αυτό που γίνεται στην Πολωνία, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία και από αυτή την οπτική γωνία αποτελεί σημαντικότατο σημείο να βρούμε ένα ορισμό ομοιογενή. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας και νομίζω ότι συμφωνούμε ιδιαίτερα με όσα ακούστηκαν εδώ. Αν δεν υπάρχουν περαιτέρω σχόλια θα ήθελα να προτείνω να καταθέσουμε μια προθεσμία 22 ε, Φεβρουαρίου για την κατάθεση τροπολογιών. Είναι σημαντικό, είναι η μόνη απόφαση που έπρεπε να λάβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, κύριο Καρόνα. Θα συναντηθούμε στις 3 ε, το απόγευμα και όπως ξέρετε θα Έχουμε την έκθεση για, την, για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ.